May I ask you to see... Σας παρακαλώ καθίστε. Please take a seat. Καθίστε παρακαλώ. Can start with the... ώστε να ξεκινήσουμε με την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βαλντής Ντομπρόσκης, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και υποψήφιο πρόεδρο για μια οικονομία που, ε, επίτροπο, συγγνώμη, για μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους. Ε, με χαρά συμπροεδρεύω με την κυρία Νικολσόνοβα. Η Επιτροπή Προπολογισμών, που είναι συνδεδεμένη ε, επιτροπή, ε, έχει εκπροσώπηση σήμερα. Πριν αρχίσει η ακρόαση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βάσει των κατευθυντηριών γραμμών για την ε, επιβεβαίωση του Επιτρόπου, που είναι παράρτημα στον κανονισμό, το Κοινοβούλιο αξιολογεί του υποψηφίου επιτρόπου βάσει των γενικότερων αρμοδιοτήτων του, την ευρωπαϊκή του δέσμευση και την προσωπική του ανεξαρτησία. Αξιολογίζουν επίση τι γνώσει για το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο και τις ε, δυνατότητες προσαρμογής τους. Πριν από την αρχή ακρόαση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και υποψήφιος επίτροπος ε, είχε απαντήσει γραπτό στις ερωτήσεις. Οι γραπτές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στα μέλη σε όλες τις γλώσσες. Τέλος, ε, παρακαλώ να σημειώσετε ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν έχει υποβάλει καμία ένσταση για την διεξαγωγή της ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τινάλη. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Ντομπρόσκη εδώ στην Ακρόαση και θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο την διαδικασία της σημερινής ακρόασης, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντομπρόσκης ε, για να κάνει μια προκαταρκτική δήλωση, η οποία θα διαρκέσει ένα τέταρτο το πολύ. Στη συνέχεια θα έχουμε 25 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές σε δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος θα είναι 7 ερωτήσεις, τις οποίες θα ρωτήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο δεύτερος γύρος, 18 ερωτήσεων, βασίζεται στη συνολική κατανομή των ερωτήσεων ε, βάσει του πολιτικών ομάδων και θα έχουμε και εκπροσώπους ε, από τους ε, μη εγγεγραμμένους. Η κάθε ερώτηση θα έχει διάρκεια πέντε λεπτών. Αρχικά θα τίθεται μία ερώτηση για ένα λεπτό, η απάντηση για δύο λεπτά και μετά μία συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό και απάντηση για ένα επιπλέον λεπτό. Μετά από αυτό, μετά από τη συζήτηση, ο κύριος Δομπρόσκης θα έχει πέντε λεπτά στο τέλος της ε, συνεδρίασης για να κάνει μια καταληκτική δήλωση και θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους τους ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο τους ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ίση εκπροσώπηση. Φυσικά υπάρχει και το σφυράκι και μπορούμε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να φροντίσετε να σκέφτεστε λίγο και το χρόνο στη διάρκεια της ερώτησής σας. Επίσης, υπάρχει διερμηνία σε όλες ε, τις ε, επίσημες γλώσσες και τις 23 ε, για την γλωσσική ποικιλομορφία. Να υπενθυμίσω βεβαίως σε όλους τους ομιλητές ότι ό,τι πουν θα μεταφράζεται. επομένω, όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος, η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχει δυνατότητα να δείτε και ε, μαγνητοσκόπηση της ακρόασης στον ίδιο ιστότοπο. Πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε, δεν κάνω λάθος. Κύριε Ντομπρόσκη, έχετε το λόγο για ένα τέταρτο για την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω σήμερα το λόγο και να σας μιλήσω για αυτά που θα πρέπει να γίνουν την επόμενη πενταετία για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Κατά τη τελευταία πενταετία, ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάστηκα στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις φορές εξελέγην Ευρωβουλευτής. Συνεπώς, θεωρώ τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι το αυτονόητο και αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας μου. Φέτος συμπληρώνονται 15 έτη από την ένταξη της Λετωνίας και 5 χρόνια από την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Ως υπουργό Οικονομικών εργάστηκα κατάπαυστα για την ένταξη της ε, χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ. Η εμπειρία που έχω αποκομίσει και από την κυβερνητική μου θητεία και από τις ευρωπαϊκές μου με να πιστεύω ότι για να πετύχουμε περισσότερα, πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερο. Και μια σταθερή Ευρώπη ε, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για την ανάπτυξη και των κρατών μελών. Ένας μέγας ε, λετωνός ποιητής, ο Ράινες, είπε ότι θα επιβιώσουν εκείνοι που αλλάζουν. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσει η οικονομία μας, ε, διατηρώντας πάντα την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τα καθήκοντά μου και να συντονίσω τις εργασίες προς μια οικονομία που να εργάζεται ε, στο συμφέρον των ε, ανθρώπων. Συνεχίζω στα αγγλικά. Βλέπουμε σήμερα τον κόσμο και δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητο την οικονομική και την κοινωνική πρόοδο που να βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες, διεθνή συνεργασία και πιο ε, ολοκληρωμένες αγορές. Ο κόσμος έχει γίνει πιο ε, πολυπολικός, πιο αβέβαιος και πιο σύγκρουσιακός. Έχουν κλιμακωθεί οι εμπορικές εντάσεις. Αυτό έχει ε, ήδη απαιτήσει ένα τίμημα από την παγκόσμια οικονομία. Στην Ευρώπη το Brexit, ιδιαίτερα το άτακτο, ε, θα προκαλέσει περαιτέρω ζημίες. Επίσης αντιμετωπίζουμε και ευρύτερε προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από αυτές. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να την μετριάσουμε και μάλιστα αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω, θα πρέπει να είμαστε ε, πρωτοπόροι στην ψηφιοποίηση και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Οι δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη και η γύραση των πληθυσμών ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις αγορές μας ε, εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Όλες αυτές οι εξελίξεις θα μετασχηματίσουν σε βάθος τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και απαιτούν τη σωστή απάντηση της δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Η ευημερία της Ευρώπης και ε, το μοντέλο μας τη κοινωνική οικονομίας τη αγορά είναι αυτά που διακυβεύονται. Θα πρέπει η οικονομία να είναι στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων. Ε, είναι αλληλένδετη η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική και η βιώσιμη. Αν με εγκρίνετε, αυτή θα είναι η βάση της εργασίας μου για την επόμενη πενταετία. Επιτρέψτε μου τώρα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά. Καταρχάς, θα, στόχο έχω να ενισχύσω την οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή που αυξάνεται η παγκόσμια ανασφάλεια. Στη συνέχεια, θα εργαστώ για να εξασφαλίσω ότι η οικονομική και η βιομηχανική μας πολιτική υποστηρίζουν το μετασχηματισμό που χρειάζεται για την οικολογία και την ψηφιακή εποχή. Οι κοινωνικές μας πολιτικές θα πρέπει να συνοδεύουν αυτούς τους μετασχηματισμούς έτσι ώστε να έχουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αξιότιμοι βουλευτές, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρή παγκοσμίω. Η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο ατού μας αφορά πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές, 22 εκατομμύρια επιχειρήσεις και ένα ΑΕΠ που υπερβαίνει τα 15-3 εκατομμύρια ευρώ. Το ευρώ είναι ένα επιτυχημένο διεθνές νόμισμα. Το δεύτερο ε, που χρησιμοποιείται για πληρωμές και παγκόσμια αποθεματικά με πρώτο μόνο το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ενισχύσει την ΟΝΕ και βεβαίως η Ευρωζώνη ε, παραμένει ανοιχτή για χώρες που θέλουν ε, να ενταχθούν και εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή όπως είναι η Βουλγαρία και η Κροατία. Χρειάζεται όμως ακόμα περισσότερη βοήθεια η οικονομία μας. Θέλω να τονίσω τη δυνατότητά μας να δρούμε ανεξάρτητα. Για να είμαστε ισχυρός και σταθερός οικονομικός παίκτη. Αυτό θα μας επιτρέψει ε, να προωθήσουμε μια διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες ε, και να αντικρούσουμε την τάση προς μια περιφερειοποίηση στον κόσμο. Θέλω ε, να πω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε την ΟΝΕ ισχυρές εθνικές οικονομίες υποστηρίζουν την οικονομική ε, κυριαρχία στην Ευρώπη. Χρειάζονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι ισχυρέ οικονομίε δημιουργούν δημοσιονομικά αποθέματα σε καλού καιρού για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα ε, σε χαλεπού όταν επιβραδύνεται η οικονομία. Αυτό είναι ο στόχο ε, των κανόνων, των δημοσιονομικών που ε, υποστηρίζουν το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκοι οι κανόνε, Θα πρέπει να του απλουστεύσουμε. Η οικονομική κυριαρχία απαιτεί η Ευρωζώνη να έχει ισχυρή δύναμη πυρός για να προλαμβάνει και να καταπολεμά τι κρίσει. Αυτό σημαίνει ένα αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ε, και ε, εργαλεία ε, δημοσιονομικά για την Ευρωζώνη. Ήδη έχουμε κάνει νομικές προτάσεις. Ε, θέλουμε επίσης να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης του επιδόματος ανεργίας. Δεν μπορούμε ε, να έχουμε οικονομική κυριαρχία χωρίς ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην περασμένη θητεία προχωρήσαμε πολύ την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Ο τραπεζικός τομέας μας είναι πολύ ε, πιο γερός τώρα από τότε που αναλάβαμε το 2014. Είναι καλύτερα κεφαλοποιημένες οι τράπεζες και πιο ανθεκτικές από πλευράς ρευστότητας. Τα ταπεινά δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα έχουν πέσει κάτω από το μισό παρόλο που παραμένουν πολύ ψηλά σε κάποιες χώρες. Τώρα απομένει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να ε, βλέπουν τις καταθέσεις τους να προστατεύονται όπου και αν ζουν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Καινοτομούν, έχουν ταλέντο και αυτό είναι πραγματικά πολύ ζωτική σημασία για την οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης. Ωστόσο, ε, πολλές φορές για να αναπτυχθούν αναγκάζονται να ξενιτευθούν. Γιατί φεύγουν λοιπόν οι πρωταθλητέ μα, οι πρωταθλητέ του μέλλοντο. Ένα λόγο είναι ότι δυσκολεύονται να βρουν τη σωστή χρηματοδότηση βάσει των κεφαλαγορών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό λόγο, τον οποίο πρέπει να αναπτύξουμε την ε, Ένωση Κεφαλαγορών. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο ταμείο για να βοηθήσει τι μικρομεσαίε να βγουν στι αγορέ. Μαζί με του συναδέλφου μου θα προτείνω μια στρατηγική για να βοηθήσω τι μικρομεσαίε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την αλλαγή των ε, συστημάτων εμπορίου. Τι επόμενε εβδομάδε θα συγκεντρώσουμε του πολιτικού διευθύνοντε στην ε, κλάδο και του καταναλωτέ για να συλλέξουμε νέε ιδέε για την ανάπτυξη των κεφαλαίων η ενίσχυση τη ευρωπαϊκή ευκυριαρχία έχει να κάνει και με την ανάληψη ευθυνών για την ενσωμάτωση και την ομοιογένεια του χρηματοοικονομικού μα κλάδου. Η υποψήφια πρόεδρο Φοντερ Λάιεν μου έχει εμπιστευτεί την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Το παίρνω πολύ σοβαρά αυτό ω καθήκον και προσβλέπω στη συνεργασία με Ευρωπαίου και διεθνεί εταίρου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, επιτήρηση και την υλοποίηση, την εφαρμογή και πέρα από τα σύνορά μας. Θα ήθελα λοιπόν επίσης ε, να δοθούν ε, ε, εποπτικές καθήκοντα για την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων και στο συντονισμό και συντονισμό σε ένα ευρωπαϊκό σώμα. Αξιότιμοι βουλευτέ. Δεύτερο στόχο θα είναι η ενίσχυση τη δημοσιονομικών, δημοκονομικών και χρηματοδοτικών πολιτικών για να ενισχύσουμε την πράσινη ε, μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Όπως ξέρετε, οι συνάδελφοί μου, Φρανς Τίμερμαντς και η Μαργκρέτ Φριστάγκερ, θα, έχουν, θα αναλάβουν ε, τη διαχείριση της ε, μετάβασης αυτής του δύο τομείους αυτούς και προσβλέπω συνεργασία μαζί του. Για να χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη προς το κλίμα, η Ευρώπη χρειάζεται μαζικές και μεγάλες επενδύσεις, τρισεκατομμύρια ευρώ τι επόμενε δεκαετίες. Θα χρειαστούμε, λοιπόν, θα χρειαστούμε και δημόσιες και δυτικέ επενδύσεις. Για να ενισχύσουμε τις δυτικές επενδύσεις, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα κανονιστικά και να δώσουμε δυνατότητε και μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Από πλευρά κανονιστική, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η πρώτη περιοχή που εφάρμοσε νόμους για την χρηματοδότηση σε βιώσιμο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε τώρα για ένα ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξη για την ταξινομία και να δούμε τι είναι βιώσιμο. Και θα πρέπει να δούμε τι πρότυπα θα βρούμε για πράσινες, ε, πράσινα ομόλογα και οικολογικέ οικολογικές πλήσει. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξουμε το σχέδιο επένδυση για την Ευρώπη. Μαζί με του συναδέλφου μου θα συστήσουμε ένα σχέδιο επενδύσεων για τη βιώσιμη Ευρώπη για ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για την επόμενη δεκαετία σε βιώσιμε επενδύσει. Μέχρι το 2025 θα θέλαμε λοιπόν το ίμιση των χρηματοδοτήσεων να αφιερωθεί στο κλίμα. Να ξέρετε βουλευτέ. η Ευρώπη έχει επί πολλές δεκαετίες υπάρξει παγκόσμιος ηγέτης σε ό,τι αφορά θέματα βιομηχανίας. Για να είμαστε λοιπόν και στο μέλλον ε, ηγετικοί θα πρέπει να αντιτηρήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεργαστώ με του συναδέλφου μα για να καταστήσουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να κατα... μπορέσει η Ευρώπη να παραμείνει στην κορυφή. Και εδώ η εμπορική πολιτική έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Μπορεί να μα βοηθήσει να προωθήσουμε του ευρύτερου στόχου μα σε ό,τι αφορά την οικονομία, την τεχνολογία, την πράσινη μετάβαση, τη βιωσιμότητα και τα εργασιακά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερο εξαγωγέας και εισαγωγέας του κόσμου. Θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ε, την περιοχή εκείνη που θα θέτει τα πρότυπα σε ό,τι αφορά το ανοιχτό και το δίκαιο ε, εμπόριο. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Αυτό έχει τεράστιο δυναμικό, για παράδειγμα, δίνοντα στου ε, καταναλωτέ μεγαλύτερη και πιο γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Θα υποβάλω λοιπόν μια νέα στρατηγική για την Ευρώπη για να καταφέρουμε ό,τι παραπάνω γίνεται από το fintech και να μπορέσουμε να είμαστε παγκόσμια ανταγωνιστικά, ανταγωνιστικοί. Εκ θα πρέπει να δούμε τους κινδύνους του θέματο του ανταγωνισμού, της και της, ε, των απειλών για την ε, χρηματονομική σταθερότητα. Παράλληλα, χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά το Libra, για παράδειγμα, και τα κρυφό νομίσματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν, αξιότιμοι βουλευτέ, να τονίσουμε ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη. Άρα, τρίτο στόχο μου θα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικέ πολιτικέ μα θα εξελιχθούν για να μπορέσουν να συνοδεύσουν αυτή τη μετάβαση. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τι ζωέ των ανθρώπων χωρί να μείνει κανεί πίσω. Θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο δράση για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Πυλών για τα κοινωνικά δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση θα υποβάλουμε ε, στοχευμένε ε, νομικέ προτάσει ε, και θα ξεκινήσουμε από ένα πλαίσιο για ελάχιστου κατώτατου μισθού. Θα πρέπει επίση να τα κοιτάξουμε αυτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η κοινωνική διάσταση ήδη έχει να κάνει με το ίμιση των συγκεκριμένων μας συστάσεων ανά χώρα. Και σκοπεύω να εστιαστώ αυτό στη μελλοντική οικονομική διαχείριση. Επίση, θα ενσωματώσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ στο εξάμεινο και στου στόχου του εξαμήνου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Στην εντολή αυτή, λοιπόν, θα ξεκινήσαμε πάλι και τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων ε, στα θέματα τη πράσινη μετάβασης και τη ψηφιακή μετάβασης είναι βασική και αυτό θα θέσει σε εφαρμογή τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επίση, ε, η συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη έχει να κάνει και με την οικονομική σύγκληση και συνοχή στι ευρωπαϊκέ περιοχέ. Ε, τα ευρωπαϊκά λοιπόν ταμεία θα μα βοηθήσουν να πετύχουμε του περιβαλλοντικού στόχου και του στόχου καινοτομία για να δώσουμε σωστή και διαβίου κατάρτιση. Και επίση θα βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε του ανθρώπου και τι περιοχέ εκείνε που θα επηρεαστούν πιο έντονα από την πράσινη μετάβαση με το νέο Ταμείο δίκαιη Μετάβαση. Ένα τελευταίο στιγμή, τώρα, επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη χωρί σωστή φορολόγηση και αυτή η Επιτροπή έχει εφαρμόσει πιο πολλέ μεταρρυθμίσει σε ό,τι αφορά την δίκαιη φορολόγηση τα τελευταία πέντε χρόνια από τα τελευταία 20 και θα συνεχίσω να επιμείνω, να επιμένω και να αγωνίζομαι προ την κατεύθυνση αυτή, ε, όπω έκανα και στην προηγούμενη θητεία, για παράδειγμα, τι προτάσει μου για τι δημόσιε τις υποχρεώσεις ε, αναφορών ε, χώρα ανά χώρα. Οι πολυεθνικές λοιπόν θα πρέπει να έχουν σωστή φορολογία, γιατί δάλλω δεν είναι δίκαια τα πράγματα σε ό,τι αφορά το φορολογικό βάρο. Αξιότιμοι βουλευτέ, ω μέλο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα εργαζόμουν σε πνεύμα συναδελφικότητα και αυτό θα συνεχιστεί. Τα τελευταία πέντε χρόνια συνεργάστηκα στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σα, με χαρά θα συνεχίσω αυτή την πολύ επικοδομητική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμο είναι πριν στο χείλο μία από τι ε, μεγαλύτερε μεταβάσει και μεταρρυθμίσεις στην ιστορία. Θα πρέπει να σχηματίσουμε λοιπόν και να δημιουργήσουμε μια οικονομία η οποία θα λειτουργεί προ όφελο του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στι ερωτήσει σα. Many thanks, Mr. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντομπρόσκη και τώρα να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους εκπροσώπους των 7 πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κάρας από το ΕΛΚ παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμη αντιπρόεδρε Ντομπρόμσκης, σας ευχαριστώ πολύ για τα σαφή εισαγωγικά σας σχόλια η ανάπτυξη, ε, οι επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις πραγματικά είναι κρίσιμα για να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους παγκόσμιους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι διαφορές της Ευρώπης. Και θα πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της αναλογικότητας. Πώς θα προσεγγίσετε αυτή την ανάγκη γενικότερα και ειδικότερα ε, σε σχέση με το πακέτο Βασιλεία 3. Επίσης, πώς θα εξασφαλίσετε καλύτερη προστασία των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά ε, τη σύναψη ε, συμφωνιών επενδυτικό μετά από τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζετε τις προτάσεις δημιουργίας μιας νέας ουδέτερης πλατφόρμας επίλυσης ε, και των διακανονισμών που δεν είναι στην ε, δικαιοδοσία ενός μεμονωμένου κράτους μέλους. Mr. Karas, ε, thank you very much on... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρας για αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά το ισότιμους άρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και τις εργασίες στον τομέα της προληπτικής νομοθεσίας. Καταρχάς, Πράγματι, αυτό το οποίο διδαχθήκαμε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είναι ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Και επομένω και οι δημοσιονομικοί κανονισμοί απαιτούν συντονισμένη απάντηση σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό είναι και αυτό το οποίο έκανε η Επιτροπή της Βασιλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής της Βασιλείας που έχουν προταθεί μέχρι τούδε και όπως βλέπουμε οι τράπεζες είναι καλύτερα κεφαλοποιημένες πλέον, υπάρχει καλύτερη ρευστότητα και λιγότερη μόχλευση. Δεσμευόμαστε ακόμα σε πολυμερείς και διεθνείς συνεργασίες σε ρυθμιστικό επίπεδο. Υπ' αυτό το πνεύμα προσεγγίζουμε λοιπόν το θέμα αυτό, προκειμένου όλοι οι βασικοί παράγοντες να εφαρμόζουν όλα τα βασικά στοιχεία του κανονισμού της Βασιλείας. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρξει σημαντική ε, συνολική αύξηση στις κεφαλακές απαιτήσει ε, και μάλιστα θα υπάρχει ε, μία διαδικασία μέχρι το 2027 θα έχουν συμπεριληφθεί τα πάντα και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα εξετάσουν τα πράγματα και θα ζητήσουν περαιτέρω ανάλυση ιδιαίτερα όσον αφορά το output και φυσικά θα υπάρξει και δημόσια διαβούλευση από αυτού. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας για την απόφαση ΑΚΜΕΑ και τη λεγόμενη ενδοκινοτική ε, διαδικασία για τις συνθήκες επενδύσεων. Βάσει της απόφασης θα πρέπει να κλείσει αυτή η διαδικασία πλέον και εξετάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον και την προστασία των επενδυτών ε, σε αυτό το πλαίσιο. Ε, συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι ο τραπεζικό μα τομέα είναι διαφορετικό με τον τομέα των ΗΠΑ και είναι διαφορετικέ και οι οικονομίε μα. Επομένω, θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά πόσον θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και θα υπάρχει ω τελεστή στήριξη και επίση ε, τον τραπεζικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση, πώ σκοπεύετε να εξασφαλίσετε ότι τα συμφέρει ε, κρατών μελών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λαμβάνονται υπόψη στο και σας. Για παράδειγμα, ε, τις νέες μεταρρυθμίσεις ε, για το πρόγραμμα στήριξης και τον Ευρωπαϊκό Έλεγχο, το Europa Για την πρώτη σας ερώτηση, κατά την εφαρμογή της Βασιλείας 3, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται εκτίμηση επιπτώσεων αυτή τη στιγμή και υπάρχει και αυτή η ευρεία δημόσια διαβούλευση προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση συγκεκριμένα για τον συντελεστή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό επεκτάθηκε στη διάρκεια αυτής της θητείας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε βεβαίως τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το συντελεστή αυτό. Όσον αφορά τις ερωτήσεις τώρα για τις σχέσεις μεταξύ ε, χωρών ευρώ και εκτός ευρώ και κυρίως ε, το δημοσιονομικό μέσο για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, οι χώρες εκτός ευρώ να υπάρχει διαθεσιμότητα ενός εργαλείου για ε, που είναι αντίστοιχο ε, και με τις χώρες ευρώ. Να είναι αντίστοιχο λοιπόν και για τις χώρες εκτός ευρώ. Ευχαριστώ. Σίλβα Περέιρα τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόσκης. Καλώς ορίσατε θα είστε αρμόδιος ε, για το συντονισμό, τη μεταρρύθμιση και τη νέα εστίαση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας, ε, κυρίως το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Χαιρετίζουμε την δέσμευσή σας να υπάρχει ισχυρότερη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική διακυβέρνηση και στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενίσχυση και της κοινωνικής διάσκετασης και κυρίως του κοινωνικού πυλώνα και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ερώτησή μου είναι εξή. Πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Μπορούμε να έχουμε και δεσμευτικές ρήτρε για να ε, προωθήσουμε τις βιώσιμες επενδύσεις και τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης όπως υπάρχουν για το έλλειμμα και το χρέος ή θα θεωρείται και πάλι ίσονο σημασία η διάσταση αυτή στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στην οικονομική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πράγματι, ο στόχος του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής μας είναι να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και όπως είπα και στην αρχή να να λάβουμε υπόψη ε, και τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα και να τα θεωρούμε ως ένα. Αυτό είναι ένας τρόπος για να εντάξουμε και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην περίληψη και των κοινωνικών θεμάτων ε, και τις συστάσεις πολιτικής. Λογικά θα υπάρχει και τακτική παρακολούθηση της προόδου για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα προωθήσουμε και θέματα συστημικά σε πολιτικές για την πράσινη μετάβαση, πράσινες επενδύσεις, κυκλική οικονομία, ε, ε, ε, αποδοτικότητα των πόρων και μετάβαση γενικότερα σε όλους τους τομείς πολιτικής και όταν θα επικεντρωνόμαστε στις εθνικές επενδύσεις θα εστιάζουμε στη βιωσιμότητα Χρησιμοποιώντα και τη στενότερη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. όσον αφορά δεσμευτικές ε, ρήτρε ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όπως γνωρίζετε υπάρχει και η διαδικασία της οικονομικής ανισορροπίας και κοιτάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε και τη βιωσιμότητα στη διαδικασία της μακροοικονομικής ανισορροπίας και κοιτάμε επίσης και θέματα στόχων μείωσης εκπομπών και σε άλλες πολιτικές όπως για παράδειγμα στην Ενεργειακή Ένωση και στις δεσμεύσεις μας να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία του Παρισιού. Επομένως όλα αυτά πρέπει να γίνουν και στο πλαίσιο άλλων πολιτικών που θα προωθήσουμε στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Μία από τις βασικότερες προκλήσεις ε, για την οικονομική διακυβέρνηση θα είναι και η απάντηση για την παρούσα οικονομική επιβράδυνση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει μεγαλύτερη ε, στήριξη στη δημοσιονομική πολιτική, να χρησιμοποιήσουμε το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε αρκετέ χώρε και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε με τον κύριο Ντράγκη και την κυρία Λαγκάρτ για την ανάγκη να υπάρχει μια δημοσιονομική πολιτική την οποία θα, η οποία θα είναι πιο υποστηρικτική και ε, συμφωνείται για την μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να υπάρχει ένας χρυσός κανόνας για τις δημόσιες επενδύσεις όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ναι, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, πράγματι, όσον αφορά τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, Ω απάντηση στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι σαφές ότι χρειάζεται απάντηση και μέσω δημοσιονομικής πολιτικής. Επομένως, ναι, συμφωνώ με αυτή τη δήλωση και Ήδη τι επόμενε μέρες θα γίνει μια συζήτηση πολιτικής και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και στο Eurogroup προκειμένου να συζητηθεί η σωστή απάντηση από πλευρά πολιτική. Όπω ε, ξέρετε, είχαμε δώσει βαρύτητα στο συνολικό δημοσιονομικό βάρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Όπως ξέρετε, βάσει των Ευρωπαϊκών Δημοσιονομικών Κανόνων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Ταμείου για να έχουμε ένα benchmark το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να έχουμε ένα περιορισμένο χρυσό κανόνα ως βάση για τον προβληματισμό μας. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει και μια ευρύτερη συνένεση για να συμφωνήσουμε για το πώς ε, θα προσαρμόσουμε και θα απλοποιήσουμε του δημοσιονομικούς μας κανόνες. Ευχαριστώ. Ο Λουίς Γκαρικάνο από την ομάδα Renew Europe. Κύριε Ντομπρόφσκε, χαίρομαι που ακούω τις απόψεις σας για το τι μέλη γενέστε. Ο Μάριο Ντράγκη είχε έρθει πριν από λίγο καιρό και ε, έδωσε 12 εβδομάδες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αυτό το χρονικό ορίζοντα. Γιατί υπάρχει εδεχόμενο νέας οικονομικής κρίσης και ε, δεν ε, έχουμε ακόμα κάνει αυτά που θα πρέπει για να αποτρέψουμε μελλοντικούς κινδύνους όπως αυτό το doom loop που είχαμε το 2011. Ε, νομίζω ότι δεν έχετε κάνει αυτά που χρειάζονται και απόδειξη είναι ότι η Τραπεζική Ένωση οπισθοδρομεί. Δεν έχουμε διείσδυση μεγαλύτερη σε άλλες χώρες, ούτε διασυνοριακό δανεισμό μεγαλύτερο. Ε, και αυτό το βλέπουμε κοιτώντα και με μονομένες τράπεζες στην Ευρώπη. Τι λείπει. Ε, σίγουρα μια κοινή εγγύηση καταθέσεων, όπως είπατε. Δεύτερον, ε, ρευστότητα, ε, εξυγίανση και ε, ισχυρά στοιχεία ενεργητικού για την Ευρωζώνη. Όλα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο ο σύμμαχός σας για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πραγματικά η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα είναι υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε δύο πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης που έχουν στηθεί και ε, λειτουργούν η ενιαία εποπτεία και η ενιαία εξυγίανση με βάση το ενιαίο εγχειρίδιο. Ε, εκρεμεί ο τρίτος πυλώνας που είναι το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Ε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού για να δούμε πώς μπορεί να, να σπάσει αυτή η εμπλοκή, το αδιέξοδο ή η πολύ αργή πρόοδος ε, στο Συμβούλιο. Αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλω να πω. Ε, ελπίζουμε στα πλαίσια αυτά να έχουμε θετικές εξελίξεις από την ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου και προσβλέπουμε και στις δικές σας προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είμαστε έτοιμοι να το διευκολύνουμε κιόλα αν χρειάζονται νέα στοιχεία για να διευκολυθούν οι συζητήσεις. Άλλα θέματα που εκκρεμούν είναι το ταμείο αυτό, το νέο για την εξυγίανση, που κάνουμε ε, πρόοδο Θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, κάποια μαξιλαράκια τα λεγόμενα έμερο για την εξηγέση των τραπεζών. Αυτό είναι ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις πρώτες ε, ε, περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε αυτή η νομοθεσία. Πραγματικά πρέπει να βρούμε μία λύση για αυτό το θέμα της ρευστότητα όταν εξηγένονται οι τράπεζες και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για την ασφάλεια των καταθέσεων, ξέρετε ε, ότι έχουμε κάνει μια πρόταση ε, για ομόλογα με εγγύηση κρατική. Δυστυχώς αυτή δεν έχει προχωρήσει στο Συμβούλιο και θα δούμε πώς μπορεί να αναζωογονηθεί αυτή η συζήτηση. Συμπροματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Ντομρόφσκης. Το πιο απογοητευτικό που έχω δει πρόσφατα ήταν η νομοθεσία κατά του ξεπλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν προχώρησαν. Ο κόσμος είναι εξωφρενών. Έχουμε δει τα LuxLeaks, τα Panama Papers, ε, διάφορα τέτοια φαινόματα, φαινόμενα συγγνώμη, ξεπλήματος και θα κάνετε πρόταση για να δημιουργηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός ε, οικονομικών πληροφοριών ε, ε, για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλήματος χρήματος στις πρώτες 100 μέρες της θητείας σας. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε από τις πιο αυστηρές διεθνώς νομοθεσίες ε, με τις σχετικές οδηγίες. Ταυτόχρονα όμως η εφαρμογή εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των κρατών μελών. Και τα πρόσφατα σκάνδαλα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δείξει ότι ε, είναι ανεπαρκής η εφαρμογή. Αυτό θα πρέπει να ε, αναλάβει κάποιο φορέα Ευρωπαϊκή Ένωση αυξημένα καθήκοντα. Ποιο θα είναι ο φορέα αυτό, μπορούμε να το δούμε στην αναθεώρηση των εποπτικών αρχών, ενδεχομένω να προσθέσουμε επιπλέον εξουσίε και αρμοδιότητε στην EBA, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, γιατί αρνήθηκαν ε, να ε, παρεύουν στο μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο ξεπλήματος στην Ευρώπη. Υπάρχει θέμα λοιπόν εκεί, αλλά πραγματικά νομίζω θα ήταν σκόπιμο να μεταφερθούν αυτές οι αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κάποιο φορέ. Ο κύριος Εκχάουτ από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντομπρόφσκη ε, που βρίσκεται εδώ μαζί μα σήμερα. Καταρχά, ε, σε ό,τι αφορά ε, την κυρία Φοντερ Λάινεν, μα υποσχέθηκε μία μελέτη για την πράσινη χρηματοδότηση και εσεί είπατε εισαγωγικά ότι ο στόχο σα θα είναι ότι θα υπάρξει μία αντίκη μετάβαση για την βιώσιμη οικονομία. Είπατε επίση ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την χρηματοδότηση και θα ψάξουμε τρόπους ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια καλή αρχή, αλλά θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου τα τρισεκατομμύρια αυτά λοιπόν να κινητοποιηθούν, τα οποία θέλουμε να δαπανηθούν τι επόμενε δεκαετίε. Θα κάνουμε λοιπόν συγκεκριμένα βήματα. Καταρχά ε, δεσμεύεστε για να βάλετε μια υποχρέωση για τη βιώσιμη ε, δέσμευση για τις τράπεζες και για τους ε, διαχειριστές πόρων και για όλους αυτούς που δίνουν χρήματα για να υπάρχει αυτή η βιώσιμη επένδυση. Και δεσμεύεστε να κάνετε πρόταση δεσμευτική τις επόμενες ε, καιρό για να υπάρχουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την άμα πράσινες επενδύσεις. Ε, επίσης δεσμεύεστε να καταπολεμήσετε τέτοιες αθέμητες επενδύσεις και τέλος δεσμεύεστε του χρόνου να εγκρίνετε μια επιπρόσθετη νομοθετική πρόταση για μια ταξινομία σε ό,τι αφορά ένα πλήρε κανονιστικό πλαίσιο για το όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων βάσει τη βιωσιμότητά σα. ευχαριστώ και περιμένω συγκεκριμένε απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματά μου αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ και όντω πολύ λεπτομερεί η ερωτήση σα. Αυτό που είναι σαφέ είναι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε φιλοδόξοι στον τομέα τη βιώσιμη χρηματοδότηση και θεωρούμε ότι αυτό είναι το κανονιστικό σκέλος της πράσινη μετάβασης. Καταρχάς, εδώ φέρω την ταξινόμηση. Γιατί ξεκινάμε του τρομερεί διαλόγου για την ταξινόμηση και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν ακόμα φέτο. Η ταξινόμηση, λοιπόν, θα αποτελέσει βάση για πολλέ περαιτέρω σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι οικολογικέ, τα πάικο labels και πολλά άλλα. Σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο και θα την επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, για μέτρα με μέτρα ε, μείωση της αλλαγής του κλίματος και όπως ξέρετε θα έχουμε και άλλα συστήματα σε ό,τι αφορά την ανταξινόμηση, για να καλύψουμε πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορών από τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει ένα fitness check σε ό,τι αφορά τις εταιρείε λοιπόν αυτές και μία, μεταρρύθμιση, και μία αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τις μη χρηματοδοτικές ε, υποχρεώσεις και τις μη χρηματοδοτικές ε, αναφορές. Θα επεκταθεί αυτό και σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και θα υπάρξει επίσης μία εναρμόνιση των υποχρεώσεων για τα άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και προφανώς αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό μας στόχο. Επίσης, καταρτίζουμε μέτρα και για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τους αριθμούς για τις ε, ε, κανονικές ε, χρηματοδοτήσει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, του αποκάλυψη των στοιχείων των επενδυτών, το EEG κτλ. Αλλά και σε πολλού άλλου τομεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τι εργασίε αυτέ. Θα επιδείξουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε 30 δεύτερα για τη συμπληρωματική σα ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κ. Άικαουτ. Όταν μίλησατε για τα πράσινα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι δεσμευτικά και βιώσιμα και θα υπάρξει τέτοια υποχρέωση αποκάλυψης στοιχείων, θα είναι δεσμευτικά δηλαδή αυτά και όχι εθραντικά. Και ύστερα μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα είναι η τράπεζα του κλίματος. Τι συζητάτε λοιπόν και τι προτείνετε, συζητάμε τις πολιτικές για την δανεισμό για την ενεργεία. Θα επιτρέψετε στην ΕΤΕΠ να μην χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, ορεκτά έργα για μερικά καύσιμα. άλλο τι νόημα έχει να λέμε ότι η ΕΤΕΠ είναι μια πράσινη τράπεζα. Απάντηση. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να σα πω ότι ένα βασικό έργο για να μετατραπεί σε πράσινη τραπέζα είναι να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στο κλίμα από 25% σε 50%. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Και σταδιακά να καταργηθεί η χρηματοδότηση τη ορεικτής ενεργείας. Αυτό συγκαταλέγεται στα μέτρα τη στρατηγική αυτή, σε ό,τι αφορά τα πράσινα ομόλογα τώρα και τα σχετικά πρότυπα. Όπω ξέρετε, ζητήσαμε από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων να μα κάνει συστάσει ε, για τα πράσινα ομόλογα και τα σχετικά πρότυπα και δημοσιεύτηκε λοιπόν η σχετική έκθεση τον Ιούνιο. Δημιουργήθηκε Έγιναν λοιπόν ε, σχετικές συστάσεις για τα πρότυπα αυτά, για οποιαδήποτε ε, εκδότη ευρωπαϊκό ή διεθνή. Θα τα υποβάλουμε αυτά λοιπόν ως πρόταση στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια τώρα θα δοθούν προτάσει, ε, θα γίνουν λεπτομερίε για όλα τα έργα που προτείνονται και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοση πράσινων ομολόγων. Ευχαριστώ από την Επιτροπή Απασχόληση και την ομάδα ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Αξιότιμο κύριε Ντομπρόφσκη. Ονειρεύεστε μια οικονομία ουδέτερη κλιματικά και για να γίνει πραγματικότητα το όνειρό σα, θέλετε να πάρετε ένα δισεκατομμύριο. Πού θα το βρείτε, δεν μα το έχετε πει πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχω την αμυδρά υποψία ότι θα τα πάρετε από το φορολογούμενο και αυτό θα έχει τεράστιε κοινωνικέ επιπτώσει. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν με επιδοτήσεις ε, θέσεις απασχόλησης. Εγώ είμαι από την περιοχή Ρουρ που παλιά ήταν η κινητήρια δύναμη ε, με τον άνθρακα και το χάλιβα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει πια άνθρακας. Έχουν πάει ε, στράφη πάρα πολλά εκατομμύρια και σήμερα είμαστε το φτωχοκομείο της Γερμανίας στην περιοχή του Ρουρ. Ε, είναι φτωχά παιδιά. Δεν λειτουργούν αυτά. Κλιματική αλλαγή Πώς θα την καταπολεμήσουμε, όχι στην Ευρώπη, ευθύνεται για το 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όποιο θέλει να σώσει το κλίμα, το κάνει στην Αφρική, την Κίνα και στον Αμαζόνιο, όχι στην Ευρώπη. Πώς θέλετε να αποτρέψετε λοιπόν ε, ολόκληρες γενιές εργαζομένων και οικογένειές τους να μην ε, θυσιαστούν στο βωμό τη αγία Γκρέτα και τη κλιματική αλλαγή. Οκ, okay. σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Καταρχάς, η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα και η Ευρώπη ε, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να την αντιμετωπίσει, γιατί το κόστος της αδράνειας θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Βεβαίως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρά αυτές τις κοινωνικές ανησυχίες όταν συζητούμε για την πράσινη μετάβαση. Και ε, αυτό ακριβώς ε, έχει υπόψη της να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μία από τις νέες προτάσεις θα είναι να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης για να συνοδεύσουμε αυτή τη μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη κλιματικά και να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες και τους πολίτες που πλήττονται περισσότερο από αυτή την πράσινη μετάβαση. Βεβαίω, ε, σαφέστατα χρειάζεται και αυτή η κοινωνική ε, διάσταση και ο κοινωνικός παράγων. Τώρα, Πώς θα επηρεάσει η πράσινη μετάβαση την ευρωπαϊκή οικονομία. Στη τελική ανάλυση μπορεί να είναι θετική επίπτωση. Ε, υπάρχουν ε, υπολογισμοί αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη δράση μας με την αδράνειά μας για τα κλιματικά, το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι γύρω στο 1% υψηλότερο αν εφαρμόσουμε αυτή τη δράση και θα αυξηθεί και κατά μισή ε, εκατοστιαία μονάδα και η απασχόληση. Άρα λοιπόν η αδράνεια είναι πιο ακριβή από τη δράση. Για το ε, Ευρωπαϊκό Σχέδιο Βιώσιμης Επένδυσης, εδώ θέλουμε να μοχλεύσουμε ιδιωτικές με βιώσιμες ε, με δημόσιες συγγνώμη, επενδύσεις, να ε, χρησιμοποιήσουμε τα ιδιωτικά κεφάλαια με βάση το σχήμα που υπάρχει ήδη για να μοχλεύσουμε τα δημόσια. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ε, το πρόγραμμα αυτό δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ε, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Τι πιστεύετε για την ηλεκτροκινητικότητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι πραγματικά ο κινητήρας ε, στη Γερμανία ε, μία στις 7 θέσεις απασχόλησης εξαρτώνται από την αυτοκιοβιχανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία αντίστοιχα. Το Πανεπιστήμιο του Έσεν, το Duisburg, έχει υπολογίσει ότι θα χαθούν 240.000 θέσεις απασχόλησης. Η Continental απολύει 20.000 ε, τα ελαστικά και οι άλλοι προμηθευτές αντίστοιχα. Ξέρουμε πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον όταν ε, βγάζουμε τα ορυκτά για τις μπαταρίες, οι οποίες είναι και δηλητηριώδεις και τοξικές. Πού θα το βρείτε το ρεύμα για την ηλεκτροκίνηση. Οκ. Για αυτό που ρωτήσατε για την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα, αυτό θα είναι τμήμα της απάντησης. Θα δούμε πώς θα οργανωθεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα ΙΟΤΑΧΗ και τα φορτηγά. Αλλά πώς θα γίνει η μείωση των εκπομπών δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν όλα από ηλεκτρικά. Μπορούμε να βελτιώσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και να έχουμε και άλλες στρατηγικές Και ε, η μείωση των εκπομπών μπορεί να έρθει και από αλλού. Και αυτό μπορεί να είναι καλό για την ευρωπαϊκή οικονομία, να χρησιμοποιούμε λιγότερη εισαγόμενη ε, ενέργεια, παραγόμενη από ορυκτά για τα αυτοκίνητα, είναι καλό ε, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο ή ακόμα και κινητήρων εσωτερικής καύσης θα πρέπει φυσικά να παράγονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήλε από την ομάδα ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και Χαίρομαι για την ε, πρότασή σας ε, για αυτό το πόστο υψηλών καθηκόντων. Χαίρομαι ε, και ως λετονός. Καταρχά τώρα, στι ερωτήσει. όσον αφορά το χαρτοφυλόκιό σα για την οικονομία που ε, λειτουργεί για του ανθρώπου, ξέρουμε ότι όταν υπάρχει ε, ανάπτυξη τη αλληλεγγύη, ε, της οικονομίας, συγγνώμη, τίθεται και θέμα αλληλεγγύη. Όπως είπατε και εσεί, μιλήσατε για τον κοινωνικό πυλώνα και πρέπει να βοηθήσουμε και τη βιωσιμότητα. Το βασικό μήνυμα βεβαίω του χαρτοφυλακίου, που δεν αποφασίστηκε από εσά, δείχνει ότι κάτι έχει αποτέλεσμα για μα και νομίζω ότι το μήνυμα είναι λίγο συγκεχημένο πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα και εμείς το θεωρούμε στο ECR πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ανάπτυξης, είμαστε βέβαια μια ομάδα του, του ε, ε, ε, στα άκρα του κέντρου, αλλά θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Ε, μία ερώτηση που έθεσε το Renew Europe θα τη συνεχίσω εγώ. Σύμφωνα με το ε, Europol, πολλά από τα εγκληματικά έσοδα δημεύονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μόνο 0,5% των ε, συναλλαγών από υποθήνους στις τράπεζες φτάνουν σε εγκληματικές και ποινικέ διαδικασίες. Υπάρχει διαφορά βέβαια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Θέματα ξεπλήματος χρήματος δεν ε, συμβαίνουν μόνο στη Βαλτική. Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες πληρώνονται και σημαντικά κονδύλια ε, από ποινές ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι γίνεται με την νομοθεσία για την πάταξη της νομοποίησης παρανόμων εσόδων. Θεωρείτε όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε τη, ε, τη συνεργασία και να είναι πιο συνεκτική η συνεργασία για τις μονάδες της αστυνομίας που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Ζήλε για τα πολύ καλά σας λόγια και για την ερώτηση. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Καταρχάς, για την ερώτηση για την οικονομία και τον τίτλο «Economy that works for people». Εγώ πιστεύω ότι η έμφαση σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Θέλουμε να εστιάσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Θέλουμε να έχουμε σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ε, ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη απλώς για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, αλλά για να έχουμε ευημερία. Ε, και επομένως πρέπει να φροντίσουμε η οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε απτά ωφέλη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας ε, για το ξέπλυμα χρήματος. Πράγματι, θίξαμε το θέμα αυτό. Η εφαρμογή των κανόνων για την νομιμοποίηση παρανόμων οδών ήταν άνηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε ξανά λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο και υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, αναθέτουμε κάποια καθήκοντα για την πάταξη του ξεπλήματος ε, στο Ευρωπαϊκό Όργανο. Έχουμε αναθέσει κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η οποία θα μπορέσει καταρχάς ε, uh, that να ζητήσει από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ερευνήσουν τυχόν ε, παραβιάσεις και ε, σε ακραίες περιπτώσεις να εγκρίνει και απόφαση που αφορά απευθείας ε, τον τραπεζικό κλάδο ή το χρηματοπιστωτικό κλάδο όταν υπάρχει παραβίαση από κάποια από αυτές τις από αυτά τα ιδρύματα. Πρέπει να δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη, αλλά περιμένουμε να έχουμε περισσότερα πράγματα για το θέμα αυτό. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει χρόνο για συμπληρωματική ερώτηση, γιατί η ερώτηση διέρχεσε πάνω από δύο λεπτά. Λυπάμαι πολύ. Ο κύριο Παπαδημούλη από την ΚΟΕ. Σύρθατε, κύριε Ντομπρόφσκη. Ο τίτλο του χαρτοφυλακίου σα είναι για μια οικονομία που λειτουργεί για του ανθρώπου. Αλλά στα 15 λεπτά που παρουσιάσατε του στόχου σα, δεν είπατε τίποτα για τι εντυνόμενες κοινωνικές ανισότητες τα τελευταία χρόνια μέσα στην Ευρώπη. Η απόσταση ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς έχει μεγαλώσει δραματικά. Αν θέλετε λοιπόν μια οικονομία που να δουλεύει για τους ανθρώπους, πείτε μου τι σκοπεύετε να αλλάξετε, με ποια μέσα, με ποια μέτρα, με ποια χρήματα θα προσπαθήσετε να σταματήσετε αυτή την εκρηκτική αύξηση των ανισοτήτων. Και το δεύτερο, από τη στιγμή που συμφωνείτε ότι χρειάζεται μια ενίσχυση των δημοσιονομικών πολιτικών για να αντιμετωπιστεί η επιβράδυνση ή και ο κίνδυνος ύφεση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πείτε μου, με ποια χρήματα θα υλοποιηθεί αυτό, όταν και ο ισχνός προϋπολογισμός που παρουσιάζει η Κομισιόν περικόπτεται από το Συμβούλιο. Uh, well, Λοιπόν, για την πρώτη σας ερώτηση, για μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους. Και πάλι θα ήθελα να τονίσω το θέμα αυτό της ε, ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους πάντες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και στη διάρκεια αυτής της Επιτροπής και θα ε, συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και στην επόμενη φοιτεία. Αν δείτε, ήδη από τώρα, στα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, σχεδόν οι μισές από τις συστάσεις μας, το 44% όλων των συστάσεων, αφορούν θέματα κοινωνικά και θέματα απασχόλησης. Και αυτή η διάσταση έχει ενισχυθεί ουσιαστικά στα τελευταία χρόνια. Αν δείτε επίσης την πρότασή μας για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνουμε και πάλι ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ με 100 δις ευρώ χρηματοδότηση προκειμένου να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν κοινωνικά ζητήματα. Αν δείτε επίσης ε, και τις προτάσεις μας σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως τη φορολόγηση, ακόμα και εκεί δίνεται έμφαση στην μείωση, για παράδειγμα, της φορολόγησης ε, των ε, χαμηλά αμοιβόμενων και μετατόπιση του φορολογικού βάρους σε άλλες βάσεις οι οποίες βοηθούν περισσότερο την ανάπτυξη μπορείτε να εξετάσετε διάφορους τομείς πολιτικής. Όσον αφορά την οικονομική επιβράδυνση, σίγουρα θα χρειαστεί μια απάντηση από πλευράς πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ένα είναι τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την οικονομική ανάπτυξη και επίσης πρέπει να δούμε και απαντήσεις ε, για την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ευελιξία στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να επιτρέψουμε περιπτώσεις ε, οικονομικής ε, ύφεσης. Συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Ντομπρόφσκης, να συμμαχίσετε με το Ευρωκοινοβούλιο εκεί όπου χρειάζεται να δράσουμε από κοινού για να σταματήσει να βάζει φρένο το Συμβούλιο σε αυτά που χρειάζονται. Γιατί ούτε αυτά που μας είπατε, ούτε αυτά που θα παρουσιάσει για τον πράσινο New Deal ο κύριος Τίμερμανς, ούτε αυτά που θα παρουσιάσει η κυρία Βεστάγκερ για την ψηφιακή μετάβαση, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με ένα προϋπολογισμό 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και επίσης είσαστε διατεθειμένος να προτείνετε ένα ευρωπαϊκό οικονομικό FBI ικανό να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το οικονομικό έγκλημα. Uh, Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, αφορά το επόμενο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κάτι πολύ ψηλότερο από το 1%. Είναι 1,2% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος που είναι 1,12% σε σχέση με το 1,3% που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στα πλαίσια του Brexit, ε, το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί και λόγω Brexit. Ε, άρα δεν θα έχουμε ουσιαστική de facto αύξηση. Είναι κάτι για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του Brexit. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ πιο φιλόδοξη ε, προσέγγιση, 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο ε, για το επόμενο πολιετέ. Αν δείτε τη συζητήσει στο Συμβούλιο, ακόμα και η ταπεινή πρόταση του 1,11% τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιε χώρε φαίνεται υπερβολική θεωρώ ότι θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να δούμε τι επιπλέον στοιχεία χρειάζονται και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στο ε, πλαίσιο του πολιτές δημοσιονομικού ταμείου, ε, πλαισίου, για παράδειγμα, στο Ταμείο Προσαρμογής. Ευχαριστώ. Η κυρία Νικόλ Σνοβατόρ για το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ. Έχουμε, Έχουμε 90 λεπτά για 18 ομιλητέ και να ξεκινήσουμε με την κυρία Βαλιτέρα από το ΕΛΚ. Ε, έχετε ένα λεπτό για να κάνετε την ερώτησή σα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε αγαπητέ Βάλτη, όπως είπατε, το ευρώ είναι επιτυχές ω νόμισμα, ωστόσο έχει και αγωνισμό. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω παραπάνω τι γίνεται με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλές επιχειρήσεις και πολλούς ανθρώπους που έχουν ε, κατά νου την κοινοτομία, τα κρυπτονομίσματα, γιατί σήμερα η σχετική νομοθεσία δημιουργεί κινδύνους και έτσι οι χώρες ε, όπως για παράδειγμα η Μάλτα εγκρίνουν δική της νομοθεσίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα είναι στη φάση που εξετάζει τις δυνατότητες. Όταν ανακοινώσατε λοιπόν τις πρωτοβουλίες ότι θα κάνετε αναθεώρηση για την υφιστάμενη νομοθεσία. Είπατε σήμερα ότι θέλετε να αναπτύξετε την νομοθεσία επ' αυτών. Πώς όμως μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό αυτών των νέων νομισμάτων, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η πρόταση του Facebook για ένα νέο νόμισμα, το Libra. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. σε ό,τι αφορά τα εικονικά νομίσματα, τα κρυπτονομίσματα, γιατί ουσιαστικά ένα νόμισμα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, μόνο ένα. Αν, αν συζητάμε λοιπόν αυτά τα κρυπτονομίσματα, όπως είπατε, ορθώς κάναμε διάφορες έρευνες και μελέτες και εξετάσαμε το κανονιστικό πλαίσιο και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στις αρχές του έτους λάβαμε και προτάσεις από τα επαπτικά ιδρύματα. Και στην παρούσα φάση καταρτίζουμε ένα, ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Αυτό το θέμα λοιπόν σίγουρα είναι πολύ επίκαιρο. Πέρσι η έρευνα είχε εστιαστεί πιο πολύ στα bitcoins και σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις της αξίας των ε, νομισμάτων αυτών προκειμένου να προστατευτεί και ο επενδυτής από τους κινδύνους. Στην παρούσα όμως φάση εξετάζουμε σοβαρά το Libra, το project αυτό δεδομένου το πόσο σημαντικέ και είναι οι εταιρείε που είναι πίσω από το Libra. Προφανώς αυτό θα μπορούσε να έχει και συστημικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την οικονομική, νομισματική σταθερότητα, την προστασία των δεδομένων, ML κτλ. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ένωση Λίμπρα να μας χορηγήσει ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τα σχέδιά τους και δεν έχουμε ακόμα λάβει τα στοιχεία αυτά. Προφανώς θα χρειαστεί ρύθμιση του Λίμπρα για να υπάρξει εποπτεία και σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο και σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδυτών και σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η συμπληρωματική ερώτηση τώρα. Oh, um, Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο, ε, λάθο έκανα. Κυρία Βαϊτέρα, έχετε συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να κάνω και μια πιο γενική ερώτηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του FinTech. Πώς μπορούμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να διατηρήσουμε την ε, χρηματοδοτική σταθερότητα και πώς θα υποστηρίξει η νέα στρατηγική FinTech τις ψηφιακές τεχνολογίες στο χρηματοδοτικό μας σύστημα. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το fintech, το σχετικό δράση, το σχετικό, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ανανεωμένο σχέδιο δράση και ήδη και στο πρώτο σχέδιο δράση ε, θέλαμε να βρούμε αυτή τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προώθηση της καινοτομία από τη μία και τη αντιμετώπιση ε, των κινδύνων από την άλλη. Μία προσέγγιση λοιπόν που εφαρμόζουμε είναι η τεχνολογική ουδετερότητα, δηλαδή εξετάζουμε τη φύση του κάθε προϊόντος και τον ενδεχόμενο κίνδυνο που δημιουργεί. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη τεχνολογία που παρέχεται. Αυτό λοιπόν αφενός. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το θέμα του ότι κοιτάζουμε τα πάντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, κοιτάμε τις πλατφόρμες crowdfunding για να δούμε ποια είναι το δυναμικό για μια ευρωπαϊκή έγκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος Ουσακόφς, για ένα λεπτό. Και σας ζητώ συγγνώμη και πάλι. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και πάλι. Επανέρχομαι ε, στο σχέδιο βιώσιμων επενδύσεων. Επανειλημμένα, το είπατε και σήμερα, λέτε ότι θέλετε να βρείτε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά φανταστικό είναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω πού θα τα βρείτε αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, υποθέτω ότι θα πρέπει να χρειαστούν ανακατατάξεις. Δεν μπορεί να είναι ένα τρισεκατομμύριο φρέσκο νέο χρήμα. Ε, ένα κλάσμα θα είναι καινούρια χρηματοδότηση και ένα κλάσμα ανακατανομή πόρων. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους για το τι ποσοστό θα είναι το καθένα. Και επίσης, τι σκοπεύετε να κάνετε απέναντι στις κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη που θα είναι αντίθετα προς την ιδέα να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για τη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Από πού να αρχίσω. Από την τελευταία ερώτηση. Ελπίζω τελικά οι κυβερνήσεις να μην αντιταχθούν. Σήμερα βλέπουμε ε, τις κυβερνήσεις να συμφωνούν με τη φιλοδοξία αυτή να κινηθούμε προς μια κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Υπάρχουν χώρες που ήδη έχουν υπογράψει ε, τη Συμφωνία των Παρισίων και στενιστεί τους στόχους μείωσης των εκπομπών. Εάν θέλεις αυτούς τους στόχους θα πρέπει να απαντήσει και το ερώτημα της χρηματοδότησης. Ελπίζω αυτό να το καταλάβει και το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά το σχέδιο βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη, εδώ ε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα υποστήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων ε, καθώς επίσης ε, και μελέτη για τα έργα που χρειάζονται. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να κινητοποιείς οικονομικούς πόρους μόνο, πρέπει να είναι και τα έργα εκείνα που θα υποστηρίξουν την μετάβαση, την οικολογική. Το ποσό, ο στόχος είναι 1,3 από το πρόγραμμα Invest EU, ε, επενδύσεις στην Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θέλει να αυξήσει το ποσοστό χρηματοδότησης για το κλίμα από 25% στο 50%. Από εκεί θα βρεθεί το ε, νέο χρήμα και από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν και τα κράτη-μέλη, ε, κρατικές επενδυτικές ε, τράπεζες, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Χρειάζεται μια συνολική καθολική προσέγγιση. Το πρώτο όμως που πρέπει να γίνει είναι ακριβώς να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την βιωσιμότητα στο πρόγραμμα Invest EU και πώς θα ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη χρηματοδότηση. Συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και πάλι ε, να σας ρωτήσω ε, για να μας δώσετε, αν όχι μια πρόβλεψη, μια εικασία ενδεχομένω. 10% ή 20%. Μαντέψτε αν δεν μπορείτε να προβλέψετε. Ποια είναι τα νέα προγράμματα, οι νέες πρωτοβουλίες που θα ήταν πρόθυμοι να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτό το νέο σχέδιο επενδύσεων. Απάντηση. Ποσοστό δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή. μίλησα για στόχους ε, δανείων της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, Αυτή είναι νέοι πόροι σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Και είναι δεκάδες δις ευρώ. Βλέπουμε 30% κλιματικό στόχο στο πρόγραμμα Invest EU. Αυτό μπορεί να διευρυνθεί και να γίνει και πιο φιλόδοξο. Επίσης, έχουμε και άλλες θηρίδες στο πρόγραμμα αυτό για δεξιότητες, μικρομεσαίες και καινοτομία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες να προωθούν πράσινη τεχνολογία, να μετεκπαιδεύουν το προσωπικό, να ε, κάνουν αυτή τη μετάβαση. Και επίσης μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δίνουν μέχρι 5% των ε, πόρων που είναι στη συνδιαχείριση ε, για το πρόγραμμα Invest EU που και αυτό θα μας βοηθήσει να μοχλεύσουμε ακριβώ πολλά νέα κονδύλια. Ε, δεν πρόκειται για να κατατάξει, τα περισσότερα θα είναι καινούρια κονδύλια. Η κυρία Αλή Ευαβέλη, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ο κατασκευαστικός ε, κλάδος είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς της οικονομίας, αλλά αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις λόγω ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας των πόρων και έλλειψη εξειδικευμένων ε, εργαζομένων. Ο κλάδος αυτός λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επίση και πολύ καλά την ψηφιοποίηση. Πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας ε, και των εσόδων. Εξού και η ερώτησή μου. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα για να υπερβούμε και την έλλειψη δυναμικού που θα ήθελε να εργαστεί στον κατασκευαστικό τομέα. Υπάρχουν επενδύσεις ε, στις διάφορες περιφέρειες ε, για κατάρτιση. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα, πράγματι αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές ανάγκες ε, σε δεξιότητες. Απ' τη μια έχουμε ένα γυράσκον εργατικό δυναμικό το οποίο πρέπει κάπως να αντικατασταθεί και επίσης υπάρχουν και ενδείξεις ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Ε, προβλέπεται για το διάστημα 2021-2025 0,5% ε, αύξηση στο εργατικό δυναμικό. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι όμως που εγκαταλείπουν τον τομέα, διότι παραδοσιακά ήταν ε, ε, ο κλάδος με πολύ μεγάλο ποσοστό αποσπεσμένων εργαζομένων. Ένα 40% λοιπόν των εργαζομένων είναι, των αποσπασμένων είναι στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό που λείπει από τον κατασκευαστικό κλάδο είναι δεξιότητες. Δεξιότητες οι οποίες ε, θα χρειαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο, θα πρέπει να αλλάξουν όμως και αυτές για να ανταποκριθούν και στις ανάγκες ε, ε κτηρίων που θα είναι οικολογικά και ενεργειακά αποδοτικά και για να υποστηρίξουμε και την ψηφιακή μετάβαση στον τομέα αυτό. Τα κράτη-μέλη εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται ε, μέσω ενός επικαιροποιημένου θεματολογίου ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ. Πιστεύουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι σημαντικός για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές στον κατασκευατικό τομέα και επομένως σκοπεύουμε να συνεργαστούμε στενά με την ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και να εστιάσουμε σε θέματα ανάπτυξης δεκτυωτήτων, εργατικό δίκαιο, επαγγελματική κατάρτιση, ασφάλεια και ε, υγεία και κινητικότητα. Ε, συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι φλέγον θέμα αυτό το Green Deal τώρα. Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να ενθαρρύνετε τους εργαζομένους στον κατασκευαστικό τομέα να συμμετέχουν στην κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη μείωση του ε, οικολογικού αποτυπώματος ε, και πώς μπορείτε να ενισχύσετε τις προδιαγραφές ε, στον κατασκευαστικό τομέα και να έχετε και στοιχεία για την ποιότητα των κατασκευών. Όλα αυτά στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επ' αυτού, όπως ε, ήδη σας ανέφερα, αλλάζουν και τα πρότυπα για τα κτίρια. Πηγαίνουμε σε παθητικά κτίρια, πιο ενεργειακά αποδοτικά και φυσικά οι κατασκευαστικές διαδικασίες ε, και οι πρακτικές, αλλά ακόμα και τα υλικά στον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να είναι αντίστοιχα αυτών των αλλαγών. Αυτά θα είναι σημαντικό ε, σκέλος ε, του Ευρωπαϊκού Green Deal, διότι όπως γνωρίζουμε, τα κτίρια είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη πηγή εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια πράσινη ενεργειακή μετάβαση εάν δεν ε, υπάρχει κάτι στον ε, τομέα των κτηρίων και δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και οι αλλαγές ε, στις προδιαγραφές για τα νέα κτίρια. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί και η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων που υπάρχουν ήδη. Η κυρία Σκίτεραλ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Ντομουράφσκης. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ιούνκερ, έχετε διευρύνει τον κοινωνικό διάλογο με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα και η σημασία του κοινωνικού διάλογου για μια αποτελεσματική και βιώσιμη αγορά εργασία είναι πραγματικά ύψης της σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη θετία ε, θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τον κοινωνικό διάλογο και τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ό,τι αφορά την εφαρμογή νομοθετικών πακέτων. Με αυτά κατά νου, λοιπόν, τι συγκεκριμένα μέσα, μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να ενισχύσετε τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει σωστή συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων όταν προτείνει νομοθετικές προτάσεις για να μην υπονομεύσει τα διαφορετικά μοντέλα της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση σε ό,τι αφορά το κοινωνικό διάλογο. Πραγματικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή έκανε ε, μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο και ήμασταν Ήμουν ένα από τα πρώτα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήμουν υπεύθυνο επίσημα για θέματα κοινωνικού διαλόγου. Σκοπεύουμε λοιπόν να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο, γιατί είναι σαφέ αυτό και αποτυπώνεται και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως βασική αρχή του κοινωνικού πυλώνα. Ως αρχή υπερθμών 8 του αριθμού πυλώνα. Επίσης, ε, το θέσαμε αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά και το εθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις ε, με ε, βασικές ε, προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου και, βασικού, και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σε ό,τι αφορά τα θέματα ανάπτυξης δυναμικού και επίσης θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση του κοινωνικού διαλόγου. Θα κοιτάξουμε και τα θέματα αυτόνομων συμφωνιών σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, γιατί και οι κοινωνικοί εταίροι εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει να ενημερώσουν τις εργασίες τους σε ό,τι αφορά την ψηφιακή εποχή και προφανώς όταν υποβάλλουμε σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, τονίζουμε διαρκώς ότι θέλουμε να σεβαστούμε τα μοντέλα συλλογικών συμβάσεων στα διάφορα κράτη-μέλη, ιδιαίτερως όποτε αυτά τα μοντέλα ε, δουλεύουν ε, πολύ αποτελεσματικά. Και αυτό θα αποτελέσει κατά την τηρια γραμμή μας, όπως άλλωστε ήταν και στο παρελθόν. Η συμπληρωματική ερώτηση τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Όπως είπατε και προηγουμένως, άλλοι μία πτυχή η οποία εδώ έχει το ρόλο της είναι και η ψηφιοποίηση. Πείτε μας λοιπόν τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε προκειμένου οι εργαζόμενοι σε νέα μοντέλα εργασίας όπως για παράδειγμα πλατφόρμες να έχουν σωστές εργασιακές συνθήκες ενώ παράλληλα να μην υπονομεύσουμε το δυναμικό ανάπτυξη των τομέων αυτών ή να μην εμποδίσουμε την ψηφιακή μετάβαση τη κοινωνία μας. Ξέρουμε ότι πολλά από τα άτομα αυτά είναι αυταπασχολούμενοι. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο είδους μηχανισμό, για παράδειγμα μέσω κοινωνικού διαλόγου, για να μπορέσουν να μας πούν, να πούν στους πολιτικούς ευθύνοντες ποιες είναι οι ανησυχίες τους στη σύγχρονη κοινωνία. Πράγματι, λέει η απάντηση η ψηφιοποίηση ενέχει νέες ευκαιρίες αλλά και καινούριου κινδύνους και προκλήσεις και οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν ένα βασικό στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν όταν θα προετοιμάσουμε το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μία από τις συνιστώσεις, μία από τις σκέψεις μας θα είναι ακριβώς η βελτίωση των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ήδη έχουμε υποβάλει διάφορες προτάσεις για τροποποίηση τη οδηγία για τι εργασιακές συνθήκες και τι ε, συστάσεις του Συμβουλίου για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Γιατί εδώ αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι το εξή. Ανεξάρτητα από τις μορφές μορφέ εργασίε, οι εργαζόμενοι, εφόσον συμβάλλουν στο κοινωνικό σύστημα, θα πρέπει να καλύπτονται από αυτό. Αυτή είναι η βασική μας αρχή που διέπει τις εργασίες μας. Κύριε κυρία Ντόμπρεφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντομπρόφσκης, στις γραπτές σας απαντήσεις παραθέσατε την κυρία Φόντερ Λάιεν. Έχει έρθει η ώρα να συμφιλειωθεί η σύγχρονη οικονομία ε, και με το κοινωνικό στοιχείο και κάνετε κάποιες προτάσεις για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και την κοινωνική διάσταση και την ενίσχυσή της. Θέλω όμως συγκεκριμένα να σας ρωτήσω, θα φέρετε νομοθετική πρόταση που να συμπεριλαμβάνει την κοινωνική στέγαση, τα μισθολογικά, τις ε, ανισότητες και τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις για τις συλλογικέ συμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και βασικός στόχος είναι να έρθει νομοθεσία έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί ε, και το κοινωνικό βαθμολόγιο πίνακας επιδόσεων και με τους 20 στόχους του κοινωνικού πυλώνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Για την κοινωνική διάσταση πρώτα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχει ενισχυθεί σημαντικά ε, τα προηγούμενα έτη. Την τελευταία διετία χρησιμοποίησαμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο ακριβώς για να βελτιώσουμε και την εφαρμογή του χάρτη ε, του πυλώνα μάλλον κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Και από το 2018 υπάρχει αυτό το βαθμολόγιο που ε, βαθμολογεί τα κράτη-μέλη ε, σχετικά όπου μπορούμε να το διευρύνουμε φυσικά. Μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό ε, όταν θα καταρτήσουμε το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τώρα, το κατά πόσο χρειάζεται νομοθεσία για να παρακολουθείτε η κοινωνική στέγη, οι ανισότητες στο εισόδημα κτλ. Μα αυτό το κάνουμε ήδη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αν θέλετε να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την ουσία της ερώτησής σας. Αλλά για να καλύψουμε την κοινωνική διάσταση και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, έχουμε αυτή την πρόθεση, όντως, και γίνεται ήδη. Κάτι άλλο σημαντικό το οποίο επίσης ενισχύσαμε τα τελευταία χρόνια, είναι η δέσμευση των κρατών μελών να συνεννοούνται με τους κοινωνικούς εταίρους, με άλλους ενδιαφερομένους. Εμείς δεν δίνουμε μόνο συστάσεις στα κράτη-μέλη, αλλά συζητούμε μαζί τους για να κατανοούμε καλύτερα το εκάστοτε πλαίσιο, τις ανάγκες και την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα. Και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο γίνεται τμήμα της συζήτησης εθνικής πολιτικής. Συμπροματική ερώτηση. Η κυρία Ντόμπρεφ. Ωραία, σταματώ εδώ στην τελευταία σας πρόταση για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αυτό δίνει και, στη, και δημοκρατική νομιμοποίηση σε όλο το εγχείρημα. Θέλετε τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν και ένα ποιοτικό και διαφανή κοινωνικό διάλογο. Συγκεκριμένα λοιπόν θα κάνετε νομοθετική πρόταση για ένα πλαίσιο, για ενημέρωση, διαβούλευση, ευρεία εκπροσώπηση έτσι ώστε η διαδικασία αυτή και κυρίως ο κοινωνικός πυλώνας να γίνει πιο διαφανής διαδικασία και πιο δημοκρατική. Απάντηση. Καταρχάς, η αρχή της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και ο ρόλος τους εν γέννη είναι κατοχυρωμένη στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο παράγωγο δίκαιο. Βεβαίως, ε, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε αν χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά όμως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οι κοινωνικοί εταίροι ήδη συμμετέχουν. Έχουμε την πρόθεση αυτό να το συνεχίσουμε de facto και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς, αλλά ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη να το πραγματοποιούν σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές συστάσεις αναχώρα που απευθύνουμε σε χώρες και τους ζητούμε να ε, συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι όταν καταρτίζονται έγγραφα σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και φυσικά ζητούμε ότι τα κράτη-μέλη να μας ενημερώνουν με ποιον τρόπο συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Η κυρία Σδανόκα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Είσαστε υποψήφιο αντιπρόεδρο για τη θέση τη οικονομία ε, η οποία λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου. Ω τώρα όμω ακούμε πολλά οικονομικά στοιχεία και δεν ακούμε αρκετά για τον άνθρωπο σε ό,τι αφορά την ακρόαση αυτή, μου δίνεται η εντύπωση ότι οι εργασίες αυτές είναι... Θα πρέπει να τις αισθάνεται κοντά του ο άνθρωπος για να αισθάνεται ότι η οικονομική κατάσταση ε, ουσιαστικά προωθεί την ε, κοινωνική ζωή. Τα κοινωνικά αυτά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη ιδιαίτερα για τη χώρα μας, την Λετωνία, αλλά και για όλες τις χώρες εκείνες όπου οι κυβερνήσεις αγνοούν το θέμα των κοινωνικών εγγύησεων και θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνολό του. Ρωτώ λοιπόν, θα δεσμευτείτε να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου για την κοινωνική διάσταση σε ό,τι αφορά όλα τα νομοθετικά μέτρα και όλες τις νομοθετικές προτάσεις σε ό,τι αφορά και αυτές ιδιαίτερως που ενδεχομένως να έχουν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Απάντηση. Κοιτάξτε. Σε ό,τι αφορά την εργασία μας για τον κοινωνικό τομέα, για τον κοινωνικό κλάδο, θα είμαστε πάρα πολύ φιλοδόξοι σε ό,τι αφορά το κοινωνικό αυτό σκέλος σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης που θα προετοιμάσουμε για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα υποβάλουμε μία αναμοφωτική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά των μισθών. Για μία νέα εγγύηση για τα παιδιά, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εγγύησης για τη νεολαία, για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ενεργείας και αυτά τα αναφέρω ως παραδείγματα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα είναι φιλόδοξη στον κοινωνικό τομέα τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ε, κοινωνικής μελέτης αντικτύπου, ήδη στην παρούσα φάση κάνουμε μελέτες αντικτύπου για όλες τις νομοθετικές μας προτάσεις, ε, σύμφωνα και με τις ε, γραμμές της καλύτερης νομοθεσίας better regulation. Και η κοινωνική διάσταση συγκαταλέγεται λοιπόν σε αυτές τις πτυχές που εξετάζονται στη μελέτη δικτύπου. Για παράδειγμα, προετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης ε, για την Ελλάδα το 2015. Τότε λοιπόν ένα από τα στοιχεία που εξετάσαμε σε ό,τι αφορά τη συνεργασία αυτή ήταν και μια κοινωνική μελέτη αντικτύπου του προγράμματος. Μια μελέτη κοινωνικού αντικτύπου όταν ε, αυτό το είχαμε κατά νου λοιπόν σε όλες μας τις επαφές με τις ελληνικές αρχές. Άρα σίγουρα αυτό θα αποτελέσει ε, μέρος της λήψης αποφάσεων. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις αυτές. Η ερώτηση ήταν ναι, απλή, ναι ή όχι. Αυτό το ναι λοιπόν που μας είπατε θα πρέπει να υποστηριχθεί και από την ε, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τους κάτω τους μισθούς, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις της κυρίας Απάντηση. Να σας πω το εξή. Φυσικά, όταν συζητάμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς, αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ θα ήθελα να βάλω ένα σταρίσκο, Μιλάμε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την, ευρωπαϊκή, για την ανεργία. Αυτό είναι μια λειτουργία της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Αυτό συμπεριλαμβάνει λοιπόν και όλες τις ε, χώρες της Ευρωζώνης, αλλά έχουμε και χώρες που δεν έχουν περιθώριο ελιγμού σε ό,τι αφορά την πολιτική για τη χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική. Άρα κοιτάμε αυτή την σταθερότητα τη χρηματοδοτική στην Ευρωζώνη. Κύριε Επίτροπε. Εδώ και χρόνια η Financial Action Task Force, Manival, και ε, ε, το δικαστήριο ότι και ΜΚΟ μπορεί να κάνουν ξεπλήμα χρήματος και να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Ο Κένεθ Βέιν αρμόδιος ε, από την ε, Μαλτέζικη κυβέρνηση για ε, τις ΔΕΚΟ και τις ΜΚΟ ζήτησε να διευρυνθεί η σχετική νομοθεσία και να καλύπτει και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μετά από πολιτικές πιέσεις αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο οι ΜΚΟ εξαιρούνται από την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η απάντηση ήταν σκέτο σκάνδαλο. Και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να θεωρούνται εγκληματίες. Με άλλα λόγια, επειδή η ΜΚΟ συνήθως είναι το τσιράκι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιους τομείς όπως είναι η μεταναστευτική πολιτική, είναι και η υπεράνω του νόμου. Θα ήθελα αυτό το θέμα να το βάλω στο γραπτό κατάλογο ερωτήσεων. Δυστυχώς κόπηκαν οι ερωτήσεις μου από τους συναδέλφους που εκπροσωπούν τις μεγάλες ομάδες εδώ της πλειοψηφίας. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα. Πρώτον, για ποιο λόγο κατά την άποψή σας ασκείται ισχυρή πολιτική πίεση να εξαιρούνται από τα νομικά πλαίσια οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μιλώ πάντα για το ξέπλυμα. Δεύτερον, δεν θα κάνω συμπληρωματική, δεν θα κάνω, εντάξει. Ε, λοιπόν, δεύτερον, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα ακολουθήσετε τις συστάσεις των αρμόδιων διεθνών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού συνεδρίου. Συγγνώμη, τελειώσατε. Είναι πάρα πολύ άδικο. Ξεπεράσατε τα δύο λεπτά, δύο λεπτά και 18. Δεν θα κάνετε συμπροματική ερώτηση. Μα το είπα μόνο μου ότι δεν θα κάνω συμπροματική ερώτηση. Και θα χρησιμοποιήσω και το σφυράκι. Μόνο απάντηση, όχι συμπροματική ερώτηση. Ναι, μα το είπα κι εγώ, κύριε Επίτροπε. Uh, Σε ό,τι αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στα πλαίσια της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Είναι γεγονός ότι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, τυπικά δεν υποχρεούνται να εντάσσονται σε αυτή την οδηγία. Και επίσης δεν είναι υπόχρεες ε, και ε, με βάση τα διεθνή πρότυπα της Financial Action Task Force. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι στο πλαίσιο του ε, EML. Η ΜΚΟ είναι πελάτες ε, κάποιων ε, άλλων φορέων, αν κάνουν τραπεζικές συναλλαγές, εάν απασχολούν δικηγόρους και λογιστές και χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίοι είναι οι υποχρεοί Παρακολουθούνται λοιπόν οι δραστηριότητες και των ΜΚΙΟΝ γιατί κάποιοι πελάτες τους ή κάποιοι ε, υπάλληλοι του είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αυτά τα στοιχεία και ε, με τη δέουσα επιμέλεια που επιβάλλεται. Αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί εξαίρεση και αφορά μόνο τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τον Ιούλιο του 2019 ε, κάναμε μια εκτίμηση κινδύνου και για τις ΜΚΟ και όντως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ε, και δεν είναι μόνο οι δικές μας ε, και της αντίστοιχης Task Force για την οικονομική ανάλυση δείχνει ότι πραγματικά θα πρέπει να χρειάζεται να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά και η ΜΚΟ. Η κυρία Ραφάλσκα για ένα λεπτό. Ζου. E, w ramach swoich e, kompetencji jest Pan odpowiedzialny Στη χαρτοφυλάκια σας είστε αρμόδιος ε, για το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και ένα από τα βασικά στοιχεία που συνιστά αυτό το πυλώνα είναι να εξασφαλίσετε ίσες ευκαιρίες για όλους. Παρά την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, ε, τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το γεγονός ότι πολλοί Ευρωπαίοι είναι στο άλλο άκρο του ψηφιακού χάσματος. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί υπολογιστέ. Σε κάποιες χώρες φτάνει και το 70% ε, και κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες πληροφορικές, ε, δεν είναι στο διαδίκτυο, ε, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι αποκλείονται και κοινωνικά και οικονομικά. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει κυρίως τους ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν προκειμένου να μειώσετε αυτό το ψηφιακό χάσμα και να μην υπάρχει ψηφιακός αποκλεισμός. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αποκλεισμού, πράγματι θα αποτελέσει σημαντικό σκέλος ε, του θεματολογίου μας για την ψηφιακή αλλαγή, διότι όταν η οικονομία μας γίνει πιο ψηφιακή, οι άνθρωποι θα χρειαστούν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες. Και αυτό είναι και τμήμα του θεματολογίου για τις δεξιότητες. Πρέπει να εξοπλίσουμε τους ανθρώπους για την ψηφιακή εποχή και επομένω χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχει σαφές έλλειμμα, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις και διάφορες έρευνες και εκτιμάται ότι περίπου 30% των ανθρώπων δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες σε κατάλληλο επίπεδο για στόχους, για στόχους απασχόλησης. Ένα 10% ε, δεν έχει καμία ψηφιακή δεξιότητα, επομένως υπάρχει σαφώς ένα ε, χάσμα δεξιοτήτων το οποίο πρέπει κάπως να συμπληρώσουμε αν θέλουμε να έχουμε μια επιτυχή ε, ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό αφορά και το εκπαιδευτικό μας σύστημα βεβαίως, αλλά αφορά επίσης και τη διαβίου μάσηση ή ε, την ε, αλλαγή δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε όλη την εργασιακή μας ζωή. Ε, στη συζήτηση για το ψηφιακό χάσμα θα ήθελα να επαναλάβω και μια ακόμα ανησυχία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ψηφιακό χάσμα. Συνθήκες εργασίας εργαζομένων στην ψηφιακή οικονομία. Ιδίω ε, καθώς συζητάμε και οικονομίε ε, στις πλατφόρμες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δράσει επί του θέματος. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, μιλήσαμε και για τη σημασία της βελτίωσης στην πρόσβαση στην ψηφιοποίηση, βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, αλλά μία ακόμα πρόκληση είναι το να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την ε, εναλλασσόμενη πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων που μπορεί να δημιουργήσει ε, αποκλεισμούς διαφόρων ειδών και αποκλεισμό φυσικά από την αγορά εργασίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για τις οικονομίες μας και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τον αποκλεισμό, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο συνδέεται στενά με τις δεξιότητες. γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να αποκλειστούν από την ε, αγορά δεξιοτήτων, γιατί δεν έχουν τις ψηφιακές ε, δεξιότητες να ε, συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Ξαναρχόμαστε λοιπόν στο θέμα του θεματολογίου για τις δεξιότητες και επίσης επαναρχόμαστε και στην εγγύηση για την νεολαία. Μία από τις κατάλληλες οδούς είναι ακριβώς το γεγονός ότι αν οι νέοι άνθρωποι δεν συμμετέχουν ούτε σε απασχόληση, ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε κατόρτιση, θα πρέπει ε, η πολιτεία να τους παρέχει εντός ε, λίγων μηνών μία από αυτές τις οδούς, γιατί αν πρόκειται για νέους ανθρώπους, τα πράγματα είναι ακόμα πιο ε, ολέθρια για την υπόλοιπη εργασιακή του ζωή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζαϊχόφσκη την ερώτησή της για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία υποψήφια επίτροπε, σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό πυλώνα. Συχνά αναφέρουμε ότι υπάρχει ο στόχο ε, μια ε, δίκαιη, εύρυθμα σα ε, αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχουν καλύτεροι κανόνε, νέοι κανόνε για του πολίτε μα. Τι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, λοιπόν, νομοθετικέ και μη νομοθετικέ, σκοπεύετε να πάρετε για το τομέα τη αγοράς εργασίας σε συνεργασία με τον Επίτροπο Σμιτ και με ποιο χρονοδιάγραμμα και πότε θα εξασφαλίσετε το δικαίωμα σε ένα δίκαιο μισθό και σε μια υγειονομική περιθάλψη θα έχουν την ίδια προτεραιότητα όπως και οι φιλόδοξοι οικονομικοί στόχοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Και καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε υπεύθυνοι και για την προπαρασκευαστική εργασία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων το 2017. Και στην παρούσα φάση καταρτίζουμε το σχέδιο δράση για την εφαρμογή του πυλώνα. Γιατί σε θέματα πρακτικής εφαρμογής διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι μη ομοιογενή σε ό,τι αφορά τα κρατημέλη, σε ό,τι αφορά του διάφορου τομεί, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση λοιπόν. Επίση, προετοιμάζουμε το σχέδιο δράση για την κοινωνικό πυλώνα. Να σα αναφέρω κάποιε συγκεκριμένε προτάσει, οι οποίε ήδη έχουν δρομολογηθεί. Κάποιες αναφέρθηκα, όπω η πρωτοβουλία για τη Λίμπρα, σε ό,τι αφορά τις δικαίου μισθού, ελάχιστου μισθού. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά, η ενίσχυση του εγγύσης και των νέων, ε, όλα αυτά για το επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, η ενημερημένη ατζέντα για τις δεξιότητες, ε, βελτιωμένες συνθήκες για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, το συζητήσαμε και αυτό, και η νέα στρατηγική για τα φύλλα. Με μέτρα για δεσμευτική διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα μισθολόγια. Όλα αυτά προφανώς θα πρέπει να τα συνοδεύσουμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να βελτιωθεί η υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει όλα αυτά να συνοδευτούν και από πόρους για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου κάνουμε πρόταση πάνω από 100 δις ευρώ για το Ευρωπαϊκό, νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο, Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Η συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το πιο ευάλωτο πληθυσμό του κοινωνιών μας, τους ε, συνταξιούχους. Μία σειρά ανθρώπων ε, στην αγορά εργασία εργάζονται σε άλλα κρατημέλη και όχι στην πατρίδα του. Και ακούω για πολλές περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και των ε, υπηρεσιών είναι τόσο χαμηλό επίπεδο που τελικά καταλήγουν σε μια μαύρη τρύπα πολλοί συνταξιούχοι γιατί παίρνουν μόνο τη συνταξή τους δύο χρόνια αφού βγουν στη σύνταξη και παραπάνω. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσετε αυτό το πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. σχετιάζεται να επιταχύνετε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος, για παράδειγμα, για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και σε ποια φάση βρίσκεται η προετοιμασία τέτοια νομοθεσία. Απάντηση. Πράγματι. Όταν εξετάζουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα συνταξιδευτικά δικαιώματα, μία πτύχη την οποία εξετάζουμε είναι η δυνατότητα μεταφορά των δικαιωμάτων αυτών, ανάλογα με την κατάσταση. Επί της αρχής, αυτό το δικαίωμα είναι ένα δικαίωμα που έχουν όσοι εργαζόμενοι μετακινούνται. Άρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην πράξη. Θα μπορούσε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας από αυτού, σε ό,τι αφορά τους ε, εργαζόμενους που βρίσκονται σε άλλο κράτο μέλο πριν συνταξιβοτηθούν σε ό,τι αφορά την κατοχήριση των δικαιωμάτων του. Όπω είπατε, σωστά η ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών, αλλά και η πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό κοινωνική Προστασία που θα μα βοηθήσει στην ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοβαρίκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υποψήφια Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Όπως σωστά τονίσατε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρίσιμες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι πάνω από 20 εκατομμύρια και απασχολούν περίπου τα 2 τρίτα των ευρωπαίων εργαζομένων. Σε κάποιο βαθμό, λοιπόν, ε, η οικονομία που λειτουργεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργεί και για τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Ε, σύμφωνα με την ε, επιστολή ανάθεσης της αποστολής σας, ε, θα πρέπει να καταρτήσετε στρατηγική για τις μικρομεσαίες. Αναφέρατε ότι ένα στοιχείο της στρατηγικής θα είναι το νέο ταμείο. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε και άλλα συγκεκριμένα στοιχεία, ας πούμε τρία μέτρα στα οποία θέλετε να βασίσετε τη στρατηγική σας για τις μικρομεσαίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση ε, και διασυνοριακή αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Είναι γεγονός ότι με τη συνάδελφο Μαργκρέτε ε, Βεστάγκερ θα συντονίζουμε το έργο αρκετών επιτρόπων για τη στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματικά είναι μια ευρεία στρατηγική η οποία καλύπτει αρκετές πτυχές. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι μία μόνο από τις πτυχές αυτές. Επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν ε, την ε, πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και το μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Να δούμε την αρχή της αναλογικότητας, πολύ σημαντική για τις ΜΜΕ, ε. το θέμα της γραφειοκρατίας. Τώρα, ειδικά για τη χρηματοδότηση και την πρόσβασή τους, ήδη έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες κατά την παρούσα θητεία, όπως είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παράγοντα υποστήριξης των μικρομεσαίων ε, σε όλες τις χορηγήσεις στο δανεισμό. Και στην ε, Ένωση των Κεφαλαιογορών προβλέπουμε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις χρηματαγορές ε, για να αναπτυχθούν ας πούμε απλούστευμένες απαιτήσει χειριδίου για πρόσβαση σε μεγαλύτερες χρηματαγορές κτλ στην επόμενη πρόταση θα δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε την ε, ε, συγχρηματοδότηση, μεικτή χρηματοδότηση μάλλον ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Να ε, δηλαδή διευκολύνουμε την πρόσβασή τους σε αυτή, να το συνδέσουμε όμως και με τους όρους και το κόστος πρόσβασής τους στις κανονικές κεφαλαίου αγορές απάντηση, μάλλον συμπληρωματική ερώτηση, συγγνώμη, ευχαριστώ για την απάντηση. Η συμπληρωματική ερώτηση έχει να κάνει με την ε, υπόθεση του ξεπλήματος ε, χρήματος και την καταπολέμηση. Το αναφέραμε. Να φύγουμε λίγο από τις απαντήσεις στις γραπτές που είδαμε και την αποστολή που σας έχει αναθέσει η Πρόεδρος. Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον εποπτικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα. Τι εννοώ. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα οργανωθούν τώρα συγκεκριμένα για να καλύπτουν αυτό το θέμα. Μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Justice, στις δικές σας υπηρεσίες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πώς θα το χειριστείτε αυτό εντός των δικών σας υπηρεσιών και πώς θέλετε να ενισχύσετε την ανταλλαγή πληροφοριών, την πληροφόρηση που μάλλον εκεί χωλαίνει περισσότερο σήμερα η κατάσταση. Ευχαριστώ. Απάντηση σε ό,τι αφορά τις ειδικέ εποπτικές αρμοδιότητες και καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ερχοληθούν σε αυτά. Ήδη έχουμε κάνει πρόταση για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Προκειμένου πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA, που θα πρέπει να ζητήσει να αναλάβουν δράση οι αρμόδιες εθνικές αρχές αν δεν αναλυφθεί αυτή η δράση, ε, τότε θα ε, επιβληθεί μια απόφαση στον ενδιαφερόμενο απευθείας. Αυτά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, αλλά νομίζω από το 2021 τίθεται σε ισχύ. Τώρα είναι ακόμα στο αποθυματικό. Σίγουρα χωράει περισσότερο συντονισμό και χρειάζεται περισσότερο συντονισμό, ανταλλαγή προφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρήση των καλών πρακτικών, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι συνεργάσιμοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές να επεμβαίνουν άμεσα. Συγγνώμη. Ε, επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, Ραντακόφσκι. Χωρίς μικρόφωνο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, πατρίδα μου, στη Σλοβακία, δημιουργούν τα δύο τρίτα Συγγνώμη, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Και πάλι λοιπόν ξεκινάω. Κύριε Ντομπρόσκης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πατρίδα μου τη Σλοβακία είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία των δύο τρίτων ε, των θέσεων εργασίας. Είναι σαφές ότι οποιοδήποτε σενάριο Brexit, εάν όντως έχουμε Brexit, θα έχει αντίκτυπο και στις αγορές ε, και φυσικά στις δουλειές αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τώρα έρχομαι στην ερώτησή μου. εσείς ε, ως ο μελλοντικός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία για όλους τους ανθρώπους, ε, σκοπεύετε, τι σκοπεύετε να κάνετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση Brexit. Και τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες αυτές τις επιχειρήσεις εάν δεν υπάρξει Brexit. Εγώ θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πιο ευάλωτες και πρέπει να προστατεύονται στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη για αυτές από ό,τι στο παρελθόν και αυτό φυσικά έχει σημασία για τις ε, μικρές χώρες όπως τη Λετωνία, την Εστονία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν ε, ιδιαίτερος για αυτές τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα κεφάλαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε μόνο 30 δευτερόλεπτα για συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ κύριε πίτροπε. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του Brexit. Το Brexit ε, σίγουρα θα προκαλέσει διαταραχές στην οικονομία, ιδιαίτερα αν έχουμε άτακτο Brexit χωρίς συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να βοηθήσει χώρες και περιφέρειες οι οποίες ε, θα πληγούν περισσότερο από αυτό το ενδεχόμενο εάν όντω ε, γίνουν τα πράγματα έτσι. Και επίσης διαθέσαμε και κάποια από τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά μέσα για στήριξη ε, χωρών και περιφερειών σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ιδιαίτερα για μικρές ε, χώρες για θέματα συνοχής και θα πρέπει να δούμε και αν θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων προκειμένου να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένους κινδύνους ή κάποια προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από τον Brexit, ιδίως αν γίνει άτακτο Brexit. Ε, πιστεύω όμως ότι ε, είναι και ευρύτερο το θέμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον, για την αναλογικότητα και όλα αυτά θα ε, συμπεριληφθούν στη στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αναπτύξουμε στην επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ε, συζητήθηκε με δύο λόγια η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, αλλά όσον αφορά τις χώρες που αναφέρεται, ε, θα ήθελα να τονίσω την ανάπτυξη των περιφερειακών κεφαλαιακών αγορών. Για παράδειγμα, υπήρχε σε αυτή τη θητεία η αγορά κεφαλαίων της Βαλτικής και θέλουμε να υποστηρίξουμε και άλλες μικρότερες χώρες για την ανάπτυξη των κεφαλαγορών τους και των περιφερειακών κεφαλαγορών. 30 δευτερόλεπτα για συμπληρωματική ερώτηση. Όσον αφορά εσάς, φαντάζομαι ότι είναι τιμή για εσάς να είστε πρωθυπουργό όταν ε, η Air ε, είχε ζημίες 250 εκατομμύρια ευρώ και 20 ε, δις κύκλο εργασιών και τώρα είναι ένας από τους καλύτερους εργοδότες. Αυτό έγινε χάρη όχι σε εσά τόσο, αλλά κάποιος από τη δική μου την πατρίδα συμμετείχε. Θα σας αναφέρω το όνομα και είμαι περήφανος ο Σλοβάκος, ε, ο οποίο εξηγίανε την ε, αεροπορική εταιρεία και ελπίζω να έχουμε και άλλου Σλοβάκου από την Ανατολική Σλοβακία εδώ στο Κοινοβούλιο. Ήθελα να θέσω μια ερώτηση, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι κάτι με ερωτηματικό στο τέλος. The next one is Miss... Επόμενος, ο κύριος Μπέλκα. Ένα λεπτό έχετε για να κάνετε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε την Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε και στο παρελθόν στο Σύμφωνο Σταθερότητα ε, και Ανάπτυξη. Προφανώ και αυτό αποτελεί ένα θεμελιώδη θέμα και θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό, ιδιαίτερω να θέσω το θέμα τη ε, ευελιξία του, του Σύμφωνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αν δεν έχει αρκετή ευελιξία η συζήτηση για τον κοινωνικό πυλώνα, η συζήτηση για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά κάποιες χώρες, είναι πολύ δύσκολη, ίσως και άσκοπη. Ρωτώ λοιπόν, ποια είναι η κόκκινη γραμμή σας σε ό,τι αφορά τη σταθερο... την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη. Γιατί ίσως να μετακινείται αυτή η γραμμή, ίσως και να μην υπάρχει όμως. Απάντηση. Επί της αρχής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μην έχουμε πολλέ κόκκινε γραμμέ και να κοιτάξουμε πιο πολύ να εργαστούμε σε ένα πνεύμα συμβιβασμού. Έτσι ε, εργάζεται και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε ό,τι αφορά το, το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη. Η προσέγγιση μα είναι η εξή: να κάνουμε την καλύτερη χρήση τη ευελιξία στα πλαίσια του συμφώνου, ωστόσο. Και τονίζουμε την προσέγγιση αυτή στη σχετική ανακοίνωση που υποβάλαμε αρχές του 2015, όπου και χρησιμοποιήσαμε κάποιες ρήτρε για τις επενδύσεις, για τις τροφωτικές μεταρρυθμίσεις, για να επιτρέψουμε στις χώρες να αποκλίνουν από τους στόχους τους, για να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές ε, και θα συνεχίσουμε στη γραμμή αυτή σε ό,τι αφορά την ε, ευέλικτη χρήση του συμφώνου. Εκ παραλλήλου, να θυμόμαστε ωστόσο ότι έχουμε και τη σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη στο σύμφωνο. Το λέει και ο τίτλος. Να κοιτάξουμε λοιπόν και την οικονομική και χρηματοδοτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα στα κρατη τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε μια τρική ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν ξέρετε ότι οι χώρε σε καλού καιρού θα πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργούν ε, αποθέματα για να μειώσουν το χρέος και για να προετοιμαστούν για εποχές ε, ε, δύσκολων οικονομικών συνθήκων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ενίσχυση της, των επενδύσεων, της οικονομίας και θα πρέπει να ζητήσουμε από τις χώρες υψηλής απόδοσης να μειώνουν το χρέος. Συμπληρωματική ερώτηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν λοιπόν κόκκινες γραμμές μας λέτε. Αλλά μία προσπάθεια κοινή για επιτεύξη συμβιβασμού. Τι λέτε λοιπόν σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι η ευελιξία του Συμφωνού Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλο ηθικό κίνδυνο και ακόμα και σε μια ένωση μεταφορών. Τι λέτε στα άτομα αυτά. Σε μια ένωση μεταβιβάσεων. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Απάντηση. Όπως σας είπα ήδη, καταρχάς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους δύο αυτούς παράγοντες γιατί προφανώς ε, χρειάζεται και η οικοδομήση, η δημιουργία εμπιστοσύνης, γιατί βάσει της εμπιστοσύνης αυτής μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον λοιπόν συμφωνούμε για ένα πλαίσιο κοινών κανόνων, θα πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κοινοί κανόνες από όλες τις χώρες. Αυτό είναι ο ηθικός κίνδυνος που αναφέρεται. Σε ό,τι αφορά το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον τώρα. Συγκεκριμένα, όπως σας είπα, θα εργαστούμε βάσει της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Συμβουλίου που υποβάλλει κάποιες ιδέες για την απλοποίηση των κανόνων του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης. Να είναι πιο απλό να εξηγηθούν οι κανόνες αυτοί και να εφαρμοστούν. Γιατί, όπως ξέρετε, στην παρούσα φάση είναι πολύ περίπλοκη. Ο κύριος Λεβαντόφσκι, ένα λεπτό για να κάνει ερώτηση. Υποψήφια Επίτροπε, ε, έχω μια ερώτηση για την προηγούμενη εμπειρία σας. Ως Πρωθυπουργό στη Λετωνία, όπου ε, διανύσατε μια σοβαρή οικονομική κρίση και επιτυχώς καταφέρατε να βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Ε, συγχαρητήρια. Έγιναν βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθόλου δημοφιλείς, αλλά αυτό έγινε ακριβώς γιατί το χρειαζόταν η χώρα, όχι λόγω εξωτερικών πιέσεων. Εδώ πώς βλέπετε αυτό το νέο ε, πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων που δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνική βοήθεια αλλά και με την οικονομική βοήθεια για χώρες που δεν εφαρμόζουν τα όσα θα όφυλα να εφαρμόζουν ε, από το ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν υπάρχει ηθικός κίνδυνος εκεί όταν επιβραβεύεις κάποιους που δεν κάνουν τα όσα ε, θα όφυλα να είχαν κάνει. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, για τις μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα υποστήριξής τους. Ε, όντως συμμετείχα και στη χάραξη και στο σχεδιασμό του προγράμματος αυτού και μπορώ να σας εξηγήσω την ε, κεντρική ιδέα. Πρώτα απ' όλα αυτό ε, το πρόγραμμα ε, διατίθεται για όλες τις χώρες, όχι μόνο για ορισμένες που ε, εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και η κεντρική ιδέα είναι ότι υποστηρίζουμε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με οικονομικά κίνητρα. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχει εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια και το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιείται ως βάση εργασίας ως ένα μέσο των χωρών της Ευρωζώνης για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, χρηματοδοτεί ε, μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές και επενδυτικές ε, σε χώρες της Ευρωζώνης και ε, σε εθελοντική βάση και σε άλλες χώρες. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα και από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης για να υποστηριχθούν οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν επευθύνουμε λοιπόν μόνο συστάσεις ανά χώρα, αλλά δίνουμε και κάποια οικονομικά κίνητρα στις χώρες αυτές για να υποστηρίξουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι καινούργια αυτή η ιδέα. Γίνονται συζητήσεις εδώ και χρόνια για τις λεγόμενες συμβατικές υποχρεώσεις ή τη μεταρρύθμιση του ίδιου του προγράμματος ε, βάσει των συζητήσεων και των όσων προκύπτουν από αυτές. Ε, συμπληρωματική ερώτηση του κύριου Λεβαντόφσκη. Για τα μέσα, για την Ευρωζώνη που αναφέρατε, θέλω να ρωτήσω. Είχαν γίνει βαρύγδουπες και περήφανες ε, δηλώσεις για ένα προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, 55 δισεκατομμύρια για την επταετία. Ε, είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο για να σταθεροποιηθεί, πιστεύετε, η Ευρωζώνη ή όχι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε προτείνει δύο πράγματα. Πρώτον, το, το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων και τώρα το συζητούμε ως δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα με μια συγκεκριμένη κλίδα ε, σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατανομή 15 με 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι για την επταετία. Μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό το ποσό μικρό, αλλά μπορούμε να το θεωρήσουμε και ως μια μαγιά έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, τώρα έχουμε πρακτικά αποτελέσματα και προτάσεις επιτάπητο. Και υπάρχει και μια δεύτερη πρόταση για τη σταθεροποίηση που κάνουμε ε, συγκεκριμένε προτάσεις για, για ε, λειτουργία σταθεροποίησης Ε, ε, υπάρχει ένα στοιχείο επιδότησης για να καλύπτει την πληρωμή των τόκων. Και εκεί είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια το ποσό. Θα δούμε πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο και πώς μπορεί να ενταχθεί και ένα σύστημα αντασφάλισης ε, των επιδομάτων ανεργίας. Επόμενος ομιλητής. Thank Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα. Κύριε Ντομπρόσχης, ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη λεγόμενη οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους, ε, θα είστε αρμόδιος ε, για τη ε, μάχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των φορολογικών παραδείσων. Η μάχη κατά των φορολογικών παραδείσων είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας και χρειάζεται άμεση δράση. Αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν είτε κοντά στη φτώχεια είτε στις παρυφές της φτώχεια και δίνονται και δισεκατομμύρια σε φορολογικούς παραδόσους που θα μπορούσαν να ε, χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, φτώχειας. Όπως είπατε και εσείς, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι φορολογική δικαιοσύνη. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν δεσμεύεστε να προτείνετε μια ευρωπαϊκή μαύρη λίστα όλων των φορολογικών παραδείσων. Καταρχάς για να δώσουμε ένα τέλος στην παράλογη πρακτική ε, του να μην συμπεριλαμβάνονται η ευρωπαϊκή φορολογική παράδοση, όπως το Λουξεμβούργο σε αυτή τη μαύρη λίστα. Και επίσης ε, ε, να σταματήσουν οι λεγόμενες γκρίζες λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται ότι προφανής φορολογική παράδοση όπως ο Παναμάς και το Τζέρζι δεν βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. η φορολογική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ε, θα συνεχίσουν να βρίσκονται υψηλά στις προτεραιότητες ε, της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Φορολογικών Παραδείσων, έχει ε, ε, δημιουργηθεί βάσει τριών κριτηρίων. Διαφάνεια, συμμόρφωση με τα κριτήρια για την ε, διάβρωση της βάσης και την μετατόπιση των κερδών και επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16 χώρες στον κατάλογο και άλλες 34 στον, στην κρίζα λίστα. Θεωρούμε ότι ο κατάλογος αυτός ε, σε γενικές γραμμές ήταν επιτυχής, διότι δεν αφορά μόνο τις χώρες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται, αλλά δίνει και κίνητρα για αλλαγές ε, σε διάλογο με τις χώρες και από τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη λίστα αυτή, άλλαξαν πάνω από 100 επιζήμια φορολογικά καθεστώτα ε, ανά τον κόσμο. Και είναι δυναμική διαδικασία της ε, ε, λίστας αυτής. Όσο ε, εξελίσσεται το φορολογικό μας πλαίσιο και εξελίσσονται και τα ζητήματα αυτά, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται και απαιτήσει. Ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, με δύο κριτήρια για την διαφάνεια ε, και τώρα έχουμε προσθέσει και νέα. Και πράγματι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει ίσα ίσα να είναι και υψηλότερα τα πρότυπα εδώ. Για παράδειγμα, όταν εφαρμόζεται η πρωτοβουλία του ΟΣΑ για την διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών, εμείς στην πρότασή μας πήγαμε πέραν των όσων ζητούσε ο ΟΣΑ. Και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω και την πρότασή μας για την κοινή φορολογική ε, βάση επιχειρήσεων, που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και κάποια από αυτά τα θέματα. Ε, συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Βίλεμσον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντομπρόσκης. Έχω εδώ ένα άρθρο που λέει ότι η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εντός της εβδομάδος θα αφαιρεθούν από τη μαύρη λίστα και την κρή λίστα των φορολογικών παραδέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ε, ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύετε σοβαρά ότι η Ελβετία, το Ντουμπάι και το Αμπου έχουν πάψει να είναι φορολογική παράδοση. Ισχύει ότι θα αφαιρεθούν οι χώρες αυτές από τη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι κάποιο κακό ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορεί στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, όπως γνωρίζετε, η προσαρμογή του καταλόγου είναι μια διαδικασία την οποία διεξάγει το Συμβούλιο και στο επόμενο Συμβούλιο θα γίνει μια συζήτηση για τις χώρες ε, του καταλόγου αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα για συγκεκριμένε αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν ή δεν θα ληφθούν από το ΕΚΟΦΕΙΝ. Να σας πω όμως ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς εφαρμόζουμε σαφώς τη μεθοδολογία μας για όλες τις χώρες και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί συγκεκριμένη βάση για το έργο των κρατών μελών και για τις αποφάσεις τους ε, κατά πάσα πιθανότητα. Ο για ένα λεπτό. <coughs> Καλημέρα σας κύριε Ντομπρόφσκης. Οι απαντήσεις σας για το κοινωνικό πυλώνα και το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι τρομακτικά αμφίσιμες. Λέτε ότι το 40% των συστάσεων είναι κοινωνικά, αλλά για την Πορτογαλία η σύσταση ήταν να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Οι ε, Πορτογάλοι έκαναν το αντίθετο και τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ε, μετά ε, θα κάνετε νομοθετική πρόταση για να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος ειλικρινά και να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία εκπρόσωποι των εργαζομένων. Στη συνέχεια, πώς θα χρηματοδοτήσετε το πράσινο deal. Ο Νίκολας Στέρν, μεγαλύτερος Άγγλος οικονομολόγος, λέει αν θέλει να κερδίσουμε τη μάχη αυτή για το κλίμα και να δημιουργήσουμε 5 εκατομμύρια ε, θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να βάλουμε το 2% του ΑΕΠ παντού. Δυστυχώς το σχέδιο επενδύσεων που προτείνεται παρά είναι ασαφές. Όσο για την τράπεζα, για το κλίμα, ε, λέτε απλώς να ε, ε, διπλασιάσει. 15 δις. 15 δις που θα τα βρει, θα κόψει από το δικό μας προπολογισμό. Αυτά δεν είναι σοβαρά ούτε στο ύψος των περιστάσεων και δεν πρόκειται να πετύχουμε για το κλίμα. Απλή ερώτηση κύριε Ντομπρόφσκης. Μπορείτε να δεσμευτείτε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι θα βρούμε νέους ίδιους πόρους, καινούριο χρήμα σε αυτό το κεφάλαιο για να φτάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεως στα 300 δις δάνεια ετησίως Ευχαριστώ απάντηση για την υλοποίηση και εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα και την κοινωνική διάσταση του κοινωνικού εξαμήνου. Ρωτήσατε κάτι για τους κατώτατους μισθούς, αν δεν απατώμε. Φέτος στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είχαμε πέντε χώρες όπου ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, ειδικό του κατώτατου μισθού. Και Είχαμε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, κατά την ε, κατάρτιση αυτών των συστάσεων για να δούμε ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και να θέσουμε ε, το, το κέντρο βάρους στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό μπορεί να είναι ε, όχι μόνο η μισθή αλλά και τα κατώτατα επιδόματα και το κατώτατο εισόδημα. σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τις επενδυτικές και τις ε, εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές διαφέρουν βέβαια. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, μετρούμε ότι χρειάζονται από 180 μέχρι 290 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2030 για να φτάσουμε στους στόχους των Παρισίων. όταν έχεις φιλόδοξους στόχους χρειάζονται και περισσότερες επενδύσεις. Τώρα το αν θα γίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Τράπεζα Κλίματος, προχωράει ταχύτατα από το σημερινό στόχο του 25% στο στόχο του 50% που όντως είναι φιλόδοξο στόχος και εμείς κάνουμε συζητήσεις και κάνουν και οι ίδιοι στο ιστορικό τους για το πώς θα φτάσουν σε αυτό το στόχο αλλά χρειάζεται από την άλλη μεριά και μια καθοδήγηση ε, ε, για τα project, τα έργα που χρηματοδοτούνται και για τις εκτιμήσεις. 15 δις ετησίως, τα δύο τρίτα μπορούν να έρθουν και από ε, εταίρους. Δηλαδή αν είναι 45 δις το χρόνο μπορούμε σε 10 χρόνια να τα έχουμε κάνει 450. Σύντομη δεύτερη ερώτησή σας γιατί η πρώτη ήταν ε, πιο μακροσκελής. Λοιπόν, ας το πάρουμε αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ε, δημιουργήσει 240 δισεκατομμύρια του χρόνου. Το, γιατί δεν τα βάζουμε στο κλίμα. Το 2008 χρειάστηκε μία εβδομάδα ε, για να έχουν πρόσβαση οι τράπεζες στο 1-3 της ΕΚΤ και καλά κάναμε και ευτυχώς. Με 240 δις μπορείτε να καταλάβετε τι θα κάνουμε στη στέγα, στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες κτλ. Αυτά τα 240 δις αντί να πάνε στην κερδοσκοπία δεν μπορούν να πάνε στο κοινό καλό και στο κοινό αυτό στόχο. Απάντησε. Εκεί φοβάμαι ότι χρειάζομαι περισσότερα στοιχεία για να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι είναι αυτό που λέτε κέρδη, ε, διανομή κερδών. Σε τι αναφέρεστε σε αυτά τα δισεκατομμύρια. Ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι θα πάει σε βοσοτική χαλάρωση 240 δισεκατομμύρια. Και, ξέρουμε ότι αυτά τα λεφτά το 80% πήγε στην κερδοσκοπία. Μα είχατε χρόνο να ρωτήσετε, λέει η Πρόεδρος. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να πω ότι είναι ανεξάρτητη και οφείλω να σέβομαι την ανεξαρτησία της, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη. Δεν θα πούμε εμεί ε, τι αποφάσει θα πάρουν για την νομισματική πολιτική. Η Κριστίν Λαγκάρτ που αναλαμβάνει τώρα ε, έχει θέσει αυτό το θέμα του πρασινίσματος και ε, των επενδύσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Και πώς θα διοχετευθούν και τα χρήματα από την ποσοτική ε, χαλάρωση. Τώρα δεν θα πει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανεξάρτητη ΕΚΤ τι να κάνει. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για τη δουλειά σας σε ό,τι αφορά τη λετωνική κρίση και στα κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τίτλος σας είναι μια οικονομία του χαρτοφυλακίου Είναι η οικονομία που λειτουργεί υπέρ του ανθρώπου. Υπέρ του ανθρώπου, λοιπόν. Θα ήθελα να προτείνω την βοήθειά μου και τη βοήθεια των συναδέλφων, αν την επιθυμείτε, σε ό,τι αφορά αυτή την πιο δύσκολη πρόκληση. Να ξεκινήσω όμως με κάτι πιο συγκεκριμένο. Στην πρότασή σας για την ε, οδηγία, για, την, ε, για τις πιστώσεις, ε, εστιαστήκατε στις δευτερογενείς αγοράς NPL και σε ό,τι αφορά τους δανειστές. Ανησυχούμε λοιπόν για την προστασία του καταναλωτή, γιατί η φυστάμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα στεγαστικά δεν ε, εξασφαλίζει η προστασία του καταναλωτή. Συμφωνείτε με αυτή την ανησυχία και με την ανησυχία για την χρηματοοικονομική σταθερότητα λόγω των στεγαστικών για παράδειγμα. Ίσως μπορείτε να μας προτείνετε τρόπους για το πώς μπορούν να καταργηθούν τα στεγαστικά από τις δευτερογενείς αγορά ή ίσως έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή. Απάντηση. Ναι, η πρόταση στην οποία αναφέρεστε είναι στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση το μη για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να μειωθούν τα επίπεδα δηλαδή τα μερίδια των ε, δανείων αυτών στι τράπεζε μα, προκειμένου οι τράπεζε να μπορούν να δανείσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και μία από τις προτάσεις ε, οι οποίες εξετάζουμε είναι πραγματικά σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στις δευτερογενείς αγορές. Εδώ. Είναι σαφές ότι και η πώληση των δανείων στη δευτερογενή αγορά δεν ε, σημαίνει ότι θα μειώνεται η προστασία του δανειζόμενου και συμφωνούμε ότι υπάρχουν βασικές αρχές για την προστασία του καταναλωτή σε ό,τι αφορά και αυτά που κατοχυρώνονται στη σχετική οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια. Από αυτή λοιπόν την άποψη, σίγουρα θα συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων για να δούμε πώς οι ευάλωτοι δανειστές μπορούν να προστατευτούν σε ό,τι αφορά. Οι δανειολήπτες λοιπόν μπορούν να προστατευτούν ε, και έχουμε και διάφορες ε, χώρες ε, όπου έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα συστήματα για την προστασία ακριβώς των ατόμων αυτών το υποστηρίζουμε λοιπόν αυτό ως σχέδιο. Θέλουμε μια αναλογική και ισορροπημένη προσέγγιση. Είναι σημαντικό ωστόσο να εξασφαλίσουμε ότι οι δανειολήπτες τελικά δεν καταλήγουν να υπερφορτώνονται. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν προσεκτική εξέταση της δανειοληπτικής ικανότητας προτού χορηγηθούν τα δάνεια και αυτό λοιπόν θα το υποβάλουμε ως πρόταση. Έχετε 50 δεύτερα για την συμπληρωματική ερώτηση. Μάλιστα. Είναι σαφή η προτεθέσει σα λοιπόν σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση και σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου Νομίζω ότι και η Ένωση των Καταναλωτών θα πρέπει να έχει σαφή ε, θέση. Σε ό,τι αφορά την προστασία λοιπόν των χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών, έγινε μια πρόταση από το Κοινοβούλιο και συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενημέρωση, την οικονομικό αλφαβητισμό των ε, καταναλωτών, ήταν σωστή η πρόταση, αλλά δεν ε, μας κάλυψε πλήρως και χρειάζεται πιο καλή προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Δεύτερη αναφορά στο βρετανικό μοντέλο. Υπάρχει η Βρετανική Αρχή για τον έλεγχο των ε, δανείων που δίνει τέτοιε υπηρεσίε προ του καταναλωτέ για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του συστήματο. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Προστασία του Καταναλωτή στι χρηματοοικονομικέ ε, συναλλαγέ θα συμπλήρωνε το σύστημα τη ενιαία αγορά στο σημείο αυτό. Μία πρόταση που ήθελα να σας πω για την προστασία των δανειοληπτών. Εισηγάγαμε παρόμοιες ε, ρήτρε σε περίπτωση που υπάρχουν δάνεια σε ε, νομίσματα σε ό,τι αφορά τι αρνητικέ δηλαδή εξέλιξει, σε ό,τι αφορά το νομίσματα σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή τώρα. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτός, αυτό ήταν και ένα από τα μοντέλα τα οποία εξετάσαμε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Το μοντέλο Twin Peaks. Να έχουμε δηλαδή μία αρχή που να εξετάζει την προστασία του καταναλωτή και την χρηματοοικονομική συμπεριφορά και την άλλη να κοιτάει τα ζητήματα προστασίας. Αυτό το μοντέλο ωστόσο δεν προκρίθηκε. Σε ό,τι αφορά τις εποπτικές αρχές, οι οποίες συστάθηκαν, Τώρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, προστασία του καταναλωτή και την ενημέρωση του καταναλωτή με το σχετικό σχέδιο δράσης μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ραφαέλα για ένα λεπτό. Και θα μιλήσω Ολλανδικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα κύριε Ντομπρόφσκη. Σε μια ισχυρή οικονομία πάει χέρι-χέρι με ίσες ευκαιρίες για όλου. ανεξάρτητα από το ε, παρελθόν του καθενό. Γιατί αν δεν μπορεί να συμμετέχει κανεί, δεν θα μπορέσει να συμμετέχει και στην οικονομική μα ευημερία. Και το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξέρουμε και εμεί εδώ και καιρό. Και Παρ' όλα αυτά, το έτος 2019 δεν έχουν ακόμα οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες όπως οι γυναίκες. Ακόμα τα άτομα με αναπηρία, ή με χρόνιες ασθένειες ε, μένουν πίσω. Οι νέοι έχουν δύσκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι εθνοτικές και σεξουαλικές μειονότητες ε, αντιμετωπίζουν διακριτική μεταχείριση και ρατσισμό. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζεται υπέρ των, του καλού όλων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ομοιογένεια. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν προκειμένου αυτές οι συγκεκριμένε ομάδες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ε, με τι βάση θα σας κρίνουμε τελικά. Σε τι βάση θα σας κρίνουμε. Απάντηση. Κοιτάξτε. Είναι μία από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που ορίζει την ε, ισότητα των ευκαιριών ως μια βασική αρχή. Και καλή για περισσότερες δράσεις για την ε, στόχευση υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Από αυτή την άποψη θα συνεχίσουμε να προωθούμε ένα σωστό εισόδημα, ενίσχυση εισοδήματος και καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για αυτούς που βρίσκονται σε τέτοιες ε, καταστάσεις και τα κράτη-μέλη φέτο έλαβαν συγκεκριμένε συστάσει αναχώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την ενίσχυση τη κοινωνική ασφάλεια και των σχετικών δικτύων κοινωνική ασφάλεια, για τη βελτίωση τη πρόσβαση στι υπηρεσίε. Και υπάρχει και χρηματοδότηση από τα Ταμεία Συνοχή και τα Διαφορετικά Ταμεία στον επόμενο προπολογισμό τη Ένωση. Έχουμε διάφορε ομάδε που εκπροσωπούνται και όπου οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από ότι αυτές ε, κατά μέσο όρο. Για παράδειγμα, οι μετανάστες ε, βλέπουμε σε ό,τι αφορά και την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και όλους αυτούς τους δείκτες ε, σημειώνουν χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με το μέσο όρο. Αντιμετωπίζουν και κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, γιατί προφανώς και αυτό έχει να κάνει με την παραγωγικότητα. Άρα στα ναι. πλαίσια της μεταναστευτικής στρατηγικής ε, εργαζόμαστε για την ε, καλή ενσωμάτωση των μεταναστών σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία, σε ό,τι αφορά το θέμα των δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά τη γρήγορη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Όλα αυτά για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αλλά όπω και να έχει η αρχή ίσων ευκαιριών υπάρχει και θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την ενισχύει. Η συμπληρωματική ερώτηση τώρα σας ευχαριστώ πολύ για την ε, απάντηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιες ομάδες στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρία. Η απασχολησιμότητα των ανθρώπων αυτών είναι 48%, 15% ενεργεία των νέων, το χάσμα μεταξύ των φύλων. 60% σε ό,τι αφορά τη μισθολογία. Θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένες πληροφορίες. Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε τα αριθμητικά αυτά στοιχεία και για να μπορέσετε πραγματικά να διευκολύνετε τις ομάδες αυτές στην αγορά εργασία. Πείτε μας συγκεκριμένα μέτρα. Αναφερθήκατε σε κάποιες ομάδες όπου θα πρέπει να βελτιωθούν τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την νεολαία, έχουμε την εγγύηση για τους νέους, μία από τις δράσεις που προτείνουμε στο σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα δύο φύλλα. Θα υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία μεταξύ άλλων θα κοιτάει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά και το μισθολογικό χάσμα. Όπως ξέρετε, η υποψηφία πρόεδρος Φοντερ Λάιεν δίνει μεγάλη σημασία σε θέματα ισότητας των φύλων και προφανώς αυτό θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ε, εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και αυτό θα είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ε, κυρία Χούμπνερ, η οποία είναι και η τελευταία ομιλήτρια, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι το ρολόι για μένα. Θα ήθελα απλώς να πω, κύριε υποψήφια την Προεδρία, νομίζω ότι η ακρόαση αυτή δείχνει σαφώς ότι έχουν γίνει πολλά σε απάντηση για την τελευταία κρίση. Φυσικά και υπάρχουν ελλείψεις, κενά, υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Ε, και ο μηχανισμός ε, για την αντιμετώπιση του κινδύνου δεν έχει ακόμα ε, ολοκληρωθεί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό και μας είπατε κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά το να επικεντρωθούμε στα διδάγματα από την προηγούμενη κρίση είναι κάτι σημαντικό. Το να δημιουργήσουμε όμως ένα ανθεκτικό, πλήρες, θεσμικό πλαίσιο πολιτικής το οποίο θα μας βοηθήσει για το μέλλον είναι κάτι άλλο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εξή, διότι ξέρουμε σε γενικέ γραμμέ ότι συμφωνούμε προς την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μου πείτε όμως ε, την προσωπική σας εκτίμηση για το πόσο καλά εξοπλισμένη θεωρείτε ότι είναι η Ευρωζώνη σήμερα προκειμένου να αντιμετωπίσει ε, τα όσα θα φέρει το μέλλον. Πώς το βλέπετε αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αφενός ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ευρωζώνη, η Οικονομική και η Νομισματική Ένωση σίγουρα είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ ε, από ό,τι ήταν πριν από την προηγούμενη κρίση, διότι πλέον έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τον ε, κύκλο για την οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση και επικεντρωνόμαστε πολύ στα κοινωνικά ζητήματα όπω συζητήσαμε σήμερα. Υπάρχει ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητα για να υποστηρίξουμε τι χώρε τη Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Υπάρχει Τραπεζική Ένωση ε, με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης ε, και το ενιαίο οδηγό και όλα αυτά έγιναν για να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχουν λοιπόν ένα σωρό εργαλεία που περιλαμβάνουν και επίσης τις ε, νομισματικές συναλλαγές τα οποία έγιναν μετά από την κρίση. Είμαστε λοιπόν σε γενικές γραμμές πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Πρέπει ακόμα να ολοκληρώσει με την ΟΝΕ. Πρέπει η Ευρωζώνη να έχει δημοσιονομικά μέσα, τα συζητήσαμε, δημοσιονομικά μέτρα για ανταγωνιστικότητα και σύγκληση, ε, Πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση, το Ταμείο Εξυγίασης Τραπεζών, το Ήρις, ε, περαιτέρω ε, τραπεζικά ζητήματα. Πρέπει η, κεφαλαια... Ε, η Ένωση Κεφαλαιαγορών επίσης να φτάσει στο τελικό της στάδιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει ακόμα να ολοκληρώσουμε και πρέπει και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν την αθεκτικότητα των οικονομικών τους χώρων. Έχουν γίνει πολλά λοιπόν, απομένουν ακόμα πολλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε για αυτό το σκοπό. Συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Χούμπνερ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο Brexit. Δεν είναι βέβαια στην επιστολή των καθηκόντων σας, αλλά ένα μεγάλο σκέλος των ευθυνών για το Brexit είναι δική σας αρμοδιότητα, ιδίω όσον αφορά την ετοιμότητα. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα υλοποιηθεί το Brexit, είναι πολύ όμως υψηλέ οι πιθανότητε. Πού θεωρείτε ότι βρισκόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για εφεδικά μέτρα όσον αφορά την προετοιμασία μας για τον Brexit και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αν μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για την προετοιμασία του ίδιου του κλάδου, των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το Brexit, προφανώς και ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε ένα άκτακτο Brexit, αλλά ξέρουμε ότι ο χρόνος πιέζει και ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ήδη πριν από αρκετό καιρό έγινε απαραίτητη αξιολόγηση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μάλλον για την ε, χρηματοπιστωτική μας ετοιμότητα και ε, το συμπέρασμα ήταν ότι χρειαζόμαστε κάποια μέτρα για να υπάρξει ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί. Ε, και για τους κεντρικούς εταίρους μας και για τα κεντρικά αποθετήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, κάποιες εξαιρέσεις για τις κεντρικές τράπεζες και φυσικά συνεργαζόμαστε και στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όσοι συμμετέχουν στις αγορές ε, θα ε, κάνουν και την απαραίτητη προετοιμασία. Θα έλεγα ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την αρχική διορία για το Brexit ε, και από αυτή την άποψη ο κλάδος εντωμεταξύ είχε και περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει και πιθανούς ε, ε, παράπλευρους κινδύνους. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο δεύτερος γύρος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις και τον υποψήφιο επίτροπο για τις απαντήσεις του. Πριν ολοκληρώσουμε την ακρόαση θα ήθελα να ζητήσω από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο και υποψήφιο επίτροπο να μας κάνει μια σύντομη ε, παρέμβαση πέντε λεπτών πριν ε, λήξει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Δαμπρόσκης. Αξιότιμες πρόεδροι, αξιότιμα μέλη, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή ε, την πλούσια ακρόαση ε, που με εμπνέει, αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θα ε, εργαστώ σαν την προς μια οικονομία που λειτουργεί ε, υπέρ των ανθρώπων. Δηλαδή θα είναι στο κέντρο οι άνθρωποι όλων των πολιτικών μας, όλοι οι Ευρωπαίοι και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε απλώς οικονομική ανάπτυξη, αλλά οικονομική ανάπτυξη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Θα συντονίζω τακτικά μαζί με κάποιους συναδέλφους την Ελίζα Φερέιρα για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, τον Τζεντιλόνι για την ε, οικονομία και άλλους ε, αρμόδιους επιτρόπους, τον Νικολά Σμιτ, και τους άλλους δύο εκτελεστικούς ε, αντιπροέδρους, ε, Βεστάγκερ και Τίμερμανς, όλες αυτές τις προσπάθειες. Όπως ε, σας είπα και εισαγωγικά, μαζί είμαστε ισχυρότεροι ενωμένοι. Δεν μπορεί μια χώρα μέλος να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Θα συνεργαστούμε λοιπόν στενά και στο μέλλον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρούσα ακρόαση. Thank you. Thank you. Ε, ευχαριστώ κύριε Ντρομπρόφσκης ε, για τις απαντήσεις σας και τις διευκρινήσεις των προθέσεών σας σε ό,τι αφορά την ευάθυση της ΟΝΕ, ε, της απόψεις σας για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαίων Χωρών καθώς επίσης και τα θέματα τα φορολογικά, του ξεπλήματος. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανησυχούν βαθύτατα και την Επιτροπή ΕΚΟΝ και τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αφήνω τώρα το μικρόφωνο στη Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ όλους. Έχω κάνει άλλες δύο ακροάσεις υποψηφίων επιτρόπων και πρέπει να σας πω ότι ήσασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι και με τον χρόνο και ε, με όλη την ακρόαση. Ε, μας διευκολύνατε ε, τα πράγματα και τελειώνουμε εγκαίρω. Θέλω να κάνω μερικά καταληκτικά σχόλια, αλλά αφού σηκώνεστε όλοι και φεύγετε δεν θα τα κάνω. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ υποψήφιοι επίτροποι και καλή σα τύχη.